with uh, uh, my Ukrainian counterpartners. Uh, let me stop here. Thank you. Well, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι όλοι κερδίσαμε. Εσείς σφιγμομετρήσατε λίγο το κοινοβούλιο αλλά και εμείς πήραμε πολλές πληροφορίες από εσά. Και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να ακούμε, να περιμένουμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Το ένα είναι βεβαίως η ενημέρωση σε σχέση με αυτήν την ε, συνάντηση. Ε, το δεύτερο θέμα είναι να εμβαθύνουμε λεπτομερία σε μερικά από τα ε, ζητήματα. Πρόκειται για μια διαρκής και σταθερή δέσμευσή μας απέναντι στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. με τις ευκαιρίες να σας ανακοινώσω για μία ακόμα φορά ότι το σημείο 8 που αφορά τη συζήτηση για την Αλβανία θα γίνει και κλεισμένον των θυρών. Το σημείο 8 για την κατάσταση στην Αλβανία. Θα το επαναλάβω βέβαια όταν θα έρθει ο κύριος Αλμπερτίνη. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσουμε ε, σύντομα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σας παρακαλώ πολύ, ηρεμήστε, ησυχάστε και καθίστε. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στην έκθεση 2010, πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010 και θα ε, εξετάσουμε τις υποβληθήσεις τροπολογίες. Πριν δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Ρία Όουμεν Ρόιτεν, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έχουν υποβληθεί 315 τροπολογίες. Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της 9ης Δεκεμβρίου εξεφράστη η ε, επιθυμία ε, να δοθεί περισσότερος χρόνος ομιλίας σε τους σκιώδεις εισηγητάς ε, λόγω του ρόλου τους. Αγαπητοί συνάδελφοι, μην με κάνετε να χτυπάω το σφυρί μου με τέτοιο βίαιο τρόπο. Σα έλεγα λοιπόν ότι έχουν υποβληθεί 315 τροπολογίε. και στη διάρκεια της συνεδριάσεως της 9 η Δεκεμβρίου εξεφράστη η επιθυμία να δοθεί μεγαλύτερος χρόνος αγόρευσης ε, εις τους σκιώδεις εισηγητάς λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό τους ρόλο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους ε, να μιλήσουν όσο γίνεται λιγότερο οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατόν. Νομίζω ότι η συγγήτρια είναι ήδη παρούσα και επομένως χωρίς ε, καμία καθυστέρηση θα δώσω άμεσα το λόγο στη συνάδελφο Ρία Όμεν Ρόιτεν. Πρόεδρε, συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα από τη θέση αυτή εδώ, από το έντρανο αυτό, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου. Πρόεδρε, σας περιμένω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τους συναδέλφους, γιατί ποτέ δεν ε, έχω δει να εκφράζεται τόσο έντονο ενδιαφέρον να υποβάλλετε τόσο πολλές τροπολογίες όσο στην έκθεση αυτή. Και σας υπόσχομαι ότι με όλους τους κοιόδης εισηγητές θα διαβουλευτώ με άριστο τρόπο για να βρω έναν καλό συμβιβασμό. Και αυτό τι σημαίνει. Υπάρχει Υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ε, υπάρχει διερμηνία προς τα αγγλικά. Ζητώ συγγνώμη από την εισηγήτρια που τη διακόπτω. Υπάρχει προφανώς κάποιο τεχνικό πρόβλημα με την διερμηνία προς τα αγγλικά. Ελήθη, πολύ ωραία. Παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ τους συναδέλφους οι οποίοι με βομβάρδισαν με τεράστιο αριθμό τροπολογιών σας υπόσχομαι ότι τις επόμενες μέρες πολύ ενδελεχώς και εντατικά θα διαβουλευτώ με τους σκιώδεις συζητητές για να βρω ένα καλό συμβιβασμό. Και ένας καλός συμβιβασμός τι θα περιλαμβάνει να παραμερίσουμε τον πιο μεγάλο ρυθμό των τροπολογιών που γίνεται. 315 τροπολογίε καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα, Πρόεδρε, και γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι σόφρον να αναφέρω ποια είναι η στάση μου έναντι των τροπολογιών, τις οποίες καθόμουν και διάβαζα χθε μέχρι τι 12.30 ώρα το βράδυ. Τρία κριτήρια θα εφαρμόσω. Πρώτο κριτήριο. Το ψήφισμα αυτό ε, έρχεται σε μια πολύ επίκαιρη στιγμή, γιατί βρισκόμαστε λίγο πριν τις κοινοβουλευτικές εκλογές εκλογέ στην Τουρκία. Και γι' αυτό, λοιπόν, Πρόεδρε, αυτό ε, καθιστά πιο έντονη την ανάγκη να τηρήσω αυστηρά τη στάση που πάντα τηρούσαμε. Να είμαστε αντικειμενικοί, κριτικοί, επικριτικοί και προς εμάς και προς την Τουρκία, αλλά και να επιλέξουμε έναν επικοδομητικό τρόπο εργασίας. Αυτό, καταρχάς, Πρόεδρε. Κατά δεύτερον, Πρόεδρε, και θα ήθελα να το επαναλάβω και προς κάποιους συναδέλφους. Διαβάζοντας τις εφημερίδες κάθε μέρα, αναφέρονται διάφορα περιστατικά τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε και τα περιστατικά αυτά από πλευρά μου δεν μπορούμε να είναι καθοριστικά για αυτά που θα γράψουμε στην έκθεση ή για την πολιτική γραμμή την οποία θα πρέπει να ορίσουμε εδώ. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα είναι ο εκδημοκρατισμός και ο εξυγχρονισμός της Τουρκίας. Και αυτό τι σημαίνει, και αυτό το θεωρώ ότι είναι πάντα ε, σημαντικό, τα κριτήρια της Κοπεχάγης να πληρούνται. Αυτά λοιπόν ως μια πρώτερη παρατήρηση. Το ψήφισμα λοιπόν το οποίο ε, υποβάλαμε κρίνει την πρόοδο της διαδικασίας μεταρρύθμισης και εξυγχρονισμού το 2010. Το ψήφισμα παράλληλα αναφέρεται στις προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν για το 2011. Αυτό τι σημαίνει, θα πρέπει να υπάρχει επικέντρωση θεωρώ, σε μια ισορροπία και στις προτεραιότητες. Και θα πρέπει να κάνουμε και να υπάρχει μια ισορροπία. Να σας πω ότι σε 8 σελίδες συνάδελφοι δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλες τις λεπτομέρειες. Πρόεδρε, αυτά λοιπόν είχα κατά νου χτες το βράδυ, τη νύχτα που καθόμουν και διάβαζα το κείμενο. Ξέρω πολύ καλά ότι σίγουρα υπάρχουν χρήσιμες προσθήκες, ότι υπάρχουν χρήσιμες ε, ε οι οποίες θα ενισχύσουν το μήνυμα. Το μήνυμα όμως, ε, όπως σας είπα, είναι το εξή. Δεν θέλουμε περιστασιακή πολιτική, θέλουμε πολιτική επικριτική, αντικειμενική και επικοδομητική. Πρόεδρε, σε κάποιους παραγράφους έχουν υποβληθεί πάρα πολλέ τροπολογίε. και νομίζω ότι και εκεί θα ήταν ενδεχομένω δυνατόν να γίνουν βελτιώσεις του κειμένου. Για παράδειγμα, παράγραφος 8 για την ελευθερία του τύπου. Παράγραφος για την ελευθερία, την ανεξιθρησκεία. 18 και 19 παράγραφοι. Και έχει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις η συνάδελφος Μποσκούρτ για τα ε, δικαιώματα των γυναικών. Και ίσως και εδώ υπάρχει ανάγκη να υπάρξει κάποια διεύρυνση της διατύπωσης. Κάποια συγκεκριμένα σημεία να αναφέρω τώρα, Πρόεδρε. Η συνάδελφος Μποσκούρτ κατά την κατάρτιση των ε, τροπολογιών σε ό,τι αφορά την επανεισδοχή. Έχει άλλωστε η ΑΜΗΝ πολύ καλύτερη θεώρηση του τι γίνεται στην Τουρκία. Αστειεύουμε, αστειεύουμε, Πρόεδρε. Από την προηγούμενη εβδομάδα μας είπαν ο Επίτροπος Μάσουμ ότι υπάρχει μια συμφωνία επί της αρχής για την επανεισδοχή, για το readmission. Και όταν θα έχουν μπει και υπογραφέ τον επόμενο μήνα, θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε την παράγραφο αυτή. Εγώ σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσω από τώρα να συμπεριλάβω τις πολύ αριθμές τροπολογίες σε ό,τι αφορά ένα συμβιβασμό. Για την Κύπρο τώρα, Πρόεδρε. Στην πρώτη συζήτηση είχα πει ότι δεν είναι σκοπός μας να κατακτήσουμε ένα ψήφισμα για την Κύπρο. Πόσο μάλλον ότι με το ψήφισμα αυτό με το ψήφισμα αυτό να ε, εμποδίσουμε τη διαδικασία διαπραγματεύσεων που θεωρώ ότι θα έχει θετικό, ε, θετική έκβαση. Ωστόσο, δεκάδες ε, τροπολογίε κατατέθηκαν για την Κύπρο και αν μου επιτρέψετε να έχω να είμαι μέτρη οφροσύνη, να πω ότι στο σημείο αυτό χρειαζόμαστε ισορροπία και πιο μεγάλη επικέντρωση. Και θέλω να σας πω ότι θεωρώ ότι το αρχικό κείμενο ως προς αυτό ήταν πολύ καλύτερο παρόλο που προτιμώ να είμαι τριόφρον γενικά. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, με κριτικό τρόπο να κοιτάξετε τις τροπολογίες σας. Πρόεδρε, πρέπει να ακολουθήσουμε την επικέντρωση της, του ψηφίσματος να σας πω ότι η νομική υπηρεσία και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου διαπίστωσαν με σαφήνεια ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, για την άμεση συμφωνία, εμπορική συμφωνία δεν πληρεί τους όρους. Άρα δεν θα υποστηρίξω ούτε τις τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Για την Αρμενία, Πρόεδρε. Δεν είχα την τιμή να μου υποβάλουν τροπολογίες για την Αρμενία. Πολλοί συνάδελφοι είχαν αυτή την τιμή. Το βλέπω σε πολλές τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί στα αγγλικά, στα γαλλικά και το καθεξής. Για την Αρμενία πάντα ήταν σαφής η στάση μου. Πάντα λοιπόν έλεγα ότι κάθε χώρα που δεν γνωρίζει την ιστορία του δεν έχει μέλλον και γι' αυτό χάρηκα όταν υπεγράφησαν τα πρωτόκολλα. Στα πρωτόκολλα λοιπόν αυτά δεν περιλαμβάνεται μόνο η ιστορική διάσταση, αλλά και μια μελλοντική διάσταση. Ένα μέλλον για τους ανθρώπους που ζουν στα σύνορα με την Αρμενία για την βελτίωση ένα καλύτερο μέλλον με συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ και εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση προκειμένου τα πρωτόκολλα το συντομότερο δυνατόν να επικυρεθούν και να εφαρμοστούν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Δεν λέω κάτι τέτοιο, δεν διατείνομαι κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ ότι αποτελεί μια πολύ καλή αρχή για μια διαδικασία συμφιλίωσης και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε και αυτό φυσικά το έχουμε ζήσει και στις ευρωπαϊκές χώρες. Πρόεδρε, θα πρέπει να έχουμε ένα σαφές μήνυμα, ένα μήνυμα το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να ασπάσετε και η μεγάλη πολιτική πλειοψηφία. Και αυτό το λέω και προς τους σοσιαλιστές, ότι το, η δική μου η ομάδα, όπου ξέρετε ότι κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη, μπορείτε να μας προκαλείτε, αλλά κάποτε καταλήξαμε σε μία δήλωση την οποία μπορούν να προσυπογράψουν και αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν με πιο γρήγορη ταχύτητα και αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν με πιο αργή ταχύτητα. Άρα, για αυτό το πολιτικό μήνυμα πριν από τις εκλογές στην Τουρκία, για το όφελος όλων των πολιτών στην Τουρκία, σας παρακαλώ, αποσύρετε τις τροπολογίες, μην ε, κάνουμε βεβαιασμένε κινήσεις και μην σπρώχνουμε υπερβολικά και τεχνητά κάποιες διαδικασίες. Πρόεδρε, θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό κείμενο, το οποίο θα ε, έχει την υποστήριξη μεγάλης βάσης στο Κοινοβούλιο και καλό και τους Κιώδης και ε, τους άλλους συναδέλφους που ξέρουν ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές οι τροπολογίες τους να τις αποσύρουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ουμεν Ρόιτεν. Όπως έλεγα και πριν, θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητά, στους οποίους μπορώ να δώσω όμως μονάχα τρία λεπτά στον καθένα. Oh, Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μιλήσω πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Ρόμεν ε, ε, ε, Ρόιτεν να ευχαριστήσω και την ίδια για τη συνεργασία και βεβαίως να συμφωνήσω και με αυτά που είπε, δηλαδή ότι πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει η προσέγγιση μας να είναι ισορροπημένη και ότι θέλει να συνεργαστεί μαζί μας για να το επιτύχουμε αυτό και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή της, να το κάνουμε και αυτό γιατί έχουμε τον ίδιο στόχο. Συμφωνώ επίσης μαζί της για το θέμα της Κύπρου. Κατανοώ ότι οι Κύπροι συνάδελφοι κυρίως μπορεί να αισθάνονται λίγο πιο παθιασμένα όσον αφορά το θέμα αυτό και βεβαίως το σεβόμαστε. Αλλά ε, μπορούμε να έχουμε μια χωριστή συζήτηση γι' αυτό. Αυτό που θέλουμε ε, είναι να υπάρχει μια αναφορά στην Κύπρο η οποία θα είναι όσο γίνεται πιο αντικειμενική ε, και να αποφύγουμε την υπερφόρτωση του κειμένου. Επίσης να πω ότι η τουρκική πλευρά ετοιμάζεται ε, να υποβάλει κάποιες προτάσεις και προς την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει να το έχουμε και αυτό ε, στο νου μας. Άκουσα ε, αυτά που αναφέρει όσον αφορά το άμεσο εμπόριο. Θέλω να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό πριν ολοκληρώσουμε την άποψή μας. Δύο ακόμα σημεία σε σχέση με τις δικές μας τροπολογίες ε, ε, σχετικά ας πούμε με την πλήρη ένταξη, σχετικά ε, με την αύξηση της ικανότητας απορρόφησης και ολοκλήρωσης. Αυτά είναι σημεία τα οποία είναι αρκετά σημαντικά. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε θέση, ούτε αλλάξαμε θέση σε σχέση με πέρσι. Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις. Πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι η πλήρης ένταξη ε, και επομένως ε, θα πρέπει να το πούμε, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις συγκεκριμένε λέξεις. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε όσον αφορά την τροπολογία αυτή. Τέλος, καταλαβαίνω ότι προσπαθεί λίγο να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου προς όλους. Δεν αναφέρθηκε σε μένα προσωπικά προς Θεού, αλλά να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τον αριθμό των τροπολογιών. Ε, πρέπει να πω ότι η ομάδα μου δεν θέλει ε, καθόλου να επηρεάσει την κοινή γνώμη ή να μπλοκάρει οποιαδήποτε διαδικασία πριν ε, και εν ώψη των, των εκλογών πρέπει να σας πω ότι υπάρχει έτσι μία ε, κούραση όσον αφορά την κοινή γνώμη της Τουρκίας για όλη αυτή τη συζήτηση ότι βρίσκεται υπό, ε, σε προενταξιακές διαδικασίες, ότι έχει μπει ε, σε τροχιά ένταξης κτλ. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χόουιτ γιατί σεβαστήκατε και το τρίλεπτο που σας έδωσα ο κύριος Λάντορφ. Και εσείς παρακαλώ αν είναι δυνατόν να μην ξεπεράσετε τα τρία λεπτά. κύριος ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τη Ρία Όμεν Ράιτον για την καλή δουλειά που έκανε και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για τις τροπολογίες δεν μπορούσα να τις διαβάσω όλες γιατί δεν μιλάω και καλά ελληνικά, καταλαβαίνετε, αλλά οι τροπολογίες αυτές ε, που διάβασα ανοίγουν μία συζήτηση την οποία έχουμε κάνει επιτυχώς ε, τα τελευταία χρόνια για το αιτιολογικό υπαριθμό, για το αιτιολογικό, την αιτιολογική σκέψη α. Γι' αυτό λοιπόν μου κάνουν εντύπωση κάποιες τροπολογίες που υποβλήθηκα. Θεωρώ ότι στην αιτιολογική σκέψη α όπως ασύσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, βρήκαμε μια διατύπωση την οποία σπάσατε μεγάλο μέρος του Κοινοβουλίου και απεικονίζει την ομοφωνία του Κοινοβουλίου ή μεγάλο, μια μεγάλη συνένεση. Αν ξανανοίξουμε τα θέματα αυτά θα ξανανοίξουμε μια πολύ βασική συζήτηση το οποίο δεν μπορεί να επιθυμούμε δεύτερον. Ναι, πρέπει να επικεντρωθούμε σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι σε κάποια ζητήματα θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι γιατί αναφέρεται, για παράδειγμα, ποιοι νόμοι αποτελούν πρόβλημα για την ελευθερία έκφρασης. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο ε, αρμόζει σε μια έκθεση όπως αυτή και δεν θα είχα πρόβλημα να συνδυαστούν αυτά ε, με τις τροπολογίες μου. Το κείμενο με τις τροπολογίες μου. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την αντικειμενική γραμμή και στάση της ε, ΡΙΑ. Το θέμα δεν είναι η επικαιρότητα η καθημερινή, ούτε το θέμα είναι η αντιδράση σε διάφορα περιστατικά. Το θέμα είναι αντικειμενικά να εκτιμήσουμε τις προσπάθειες που καταβέλει η Τουρκία για να κάνει εξυγχρονισμό. Και βλέπουμε και μια επικριτική στάση σε ό,τι αφορά και αυτό φαίνεται και στις τροπολογίες που υπέβαλε η ομάδα μου σε ό,τι αφορά τα κάποια θεμελιώδη δικαιώματα, ελευθερία έκφραση, συνάθρησης και του καθεξής δεν αποτυπώνονται. Και θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να κάνει πολλά ακόμα η Τουρκία σε ό,τι αφορά το πρωτοκριτήριο κοπενχάγης. Να σας πω ότι πολλή συζήτηση έγινε για αυτό που στα αγγλικά ονομάζεται absorption capacity, integration capacity, ίσως όταν είναι καλύτερα να το πούμε, την ικανότητα δηλαδή ε, απορρόφησης. Είναι πιο σωστό αυτό σύμφωνα με τα κριτήρια της Κοπενχάγης, γιατί αναφέρεται ότι θα πρέπει να προωθείται η δυναμική των διαβρύνσεων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι θεμητό να προωθεί τη διαδικασία ενσωματώσης η ε, ΡΙΑ. Πρέπει να σας πω ότι κάποιες ε, τροπολογίες είναι πολύ περιαξενές. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, ε πολιτική δύναμη στην Τουρκία. Εγώ ήμουν μέρος, συμμετείχα στο στρατό, αλλά Πραγματικά τι να σας πω, αυτή η τροπολογία παριθμών 151 νομίζω ότι είναι πολύ περίεργη. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ και εσάς ε, γιατί είσαστε σύντομος. Φλότρ, τρία λεπτά. Φλότρ, τρία λεπτά. Ναι, ε, ε, ήμουν λίγο στον κόσμο μου, αλλά είχε και την Τουρκία ο κόσμος μου. Λοιπόν, 315 τροπολογίε βεβαίω ε, είναι πάρα πολλέ, αλλά κοιτάζοντά τι ε, ε, είναι λίγες αυτές οι οποίες αντιτίθενται στην κεντρική γραμμή της έκθεσης τη κυρίας Όμεν Ρόιτεν, που νομίζω ότι την συμφωνούν οι περισσότερε πολιτικές ομάδες με τη γραμμή της κυρίας Ρόιτεν υπάρχουν κάποιες ε, διορθώσεις ε, φραστικές και κάποιες ε, άλλες οι οποίες εμπλουτίζουν ή αποσαφηνίζουν κάποια στοιχεία τα οποία υπάρχουν ήδη στην έκθεση. Ε, νομίζω ότι από αυτόν δεν θα υπάρχει καμία δυσκολία και η κυρία δεν θα μπορέσει να τις ε, δεχτεί. Με τους σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους έχουμε πολλές τροπολογίες οι οποίες είτε υπογραμμίζουν τα, διακυβέρματα τα διακυβεύματα που αφορούν την ελευθεροτυπία, την ε, ελευθερία έκφραση, τα δικαιώματα των γυναικών, ακολουθούν δηλαδή την γραμμή την οποία είχα ζητήσει και από την πρώτη συζήτηση, δηλαδή να έχουμε μία αντικειμενική θετική έκθεση αφενός να επιβραβεύουμε ε, τα θετικά αφετέρου όμως να υπογραμμίζουμε και τα αρνητικά. Όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις νομίζω ότι μπορούμε λίγο ε, να διαφοροποιηθούμε. Δηλαδή είναι γεγονός ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία σιγά σιγά παίρνει όλο και μεγαλύτερη θέση ε, στον διεθνή ορίζοντα Όσον αφορά την παράγραφο 39, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να προσέξουμε λίγο, να διορθώσουμε. Όσον αφορά την Κύπρο, εγώ θα ήμουν ικανοποιημένη εάν μπορούσαμε να ξαναβρούμε τις ισορροπίες τις οποίες είχαμε βρει στην τελευταία έκθεση, γιατί αυτές οι ισορροπίες επιτρέπουν, θα μας επιτρέψουν μάλλον να μην ε, φορτώσουμε στην πλάτη της Τουρκίας ε, στοιχεία τα οποία ενδεχομένως αποτελούν και δικές μας αδυναμίες ε, γιατί στην ουσία το Κοινοβούλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το 2004 δεν κατάφερε να πει κάτι ουσιαστικό και σοβαρό για την Κύπρο. Επομένως να μην τα φορτώσουμε όλα στην πλάτη της Τουρκίας. Ε, ίδιο επιχείρημα και για την ένταξη. Θα πρέπει ε, αυτή η προοπτική να είναι μια διαδικασία open-ended ε, και από την άλλη πλευρά να πούμε ότι διαπραγματευόμαστε όχι για τη διαπραγμάτευση αλλά διαπραγματευόμαστε για την ένταξη. Τέλος, κατέθεσα μια τροπολογία για τα κεφάλαια που κατά την άποψή μου καταδεικνύει τον, ε, ε, την ελάχιστα ισορροπημένη και ε, υπεύθυνη πολιτική που ασκούμε. Λέμε ότι τα κριτήρια της Κοπεχάγης είναι αποφασιστικά, αλλά δεν μπορούμε ε, να ανοίξουμε τα δύο κεφάλαια τα οποία αφορούν τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα που αφορούν ε, τις ε, ελευθερίες. Δηλαδή, εάν δεν ανοίξουμε τα κεφάλαια αυτά, η στάση μας, τι να σας πω, θα είναι ανόητη τρία λεπτά. Μην το ξεπεράσετε το uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα αναγνωρίζω ότι στο Κοινοβούλιο και σε κάθε πολιτική ομάδα υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για το όλο ζήτημα της προσχώρησης της Κύπρου, λέει ο μιλητής, και στη δική μου την ομάδα. Η Βρετανική κυβέρνηση και πολλά μέλη της ομάδας μας βέβαια υποστήριζαν ε, την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ε, ήθελα να σχολιάσω τρεις πτυχές. Πρώτα απ' όλα. Σε ό,τι αφορά το 1915 Υπάρχουν βουλευτές που θέλουν να μιλήσουν για γενοκτονία των Αρμενίων και έχουν καταθέσει τροπολογίες. Στόχος σου είναι απομόνωση και προσβολή της Τουρκίας σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή όπου η κατάσταση είναι πάρα πολύ λεπτή για να μην πω και επικίνδυνη. Στην Τουρκία αυτό γίνεται αντιληπτό ως μια υπολογισμένη προσβολή. Η τουρκική κυβέρνηση έχει προτείνει έχει προσφέρει στις αρμενικές αρχές τη δημιουργία μιας κοινή επιτροπής που θα μελετήσει την ιστορία αυτής της αμφιλεγόμενης περίοδου για το 1915. Και δυστυχώς η Αρμενία δεν αντέδρασε θετικά, δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρωτοβουλία. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι και θέλουν να παρα, ουσιαστικά να αποστασιοποιήσουν ή να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη και να προσβάλλουν ε, δεν κάνουν σωστά και εμείς πρέπει αυτό να το αποφύγουμε πάση Τώρα για το Κυπριακό και πάλι αναγνωρίζω ε, πόσο βαθιά αισθήματα έχουν οι φίλοι μου από την Ελλάδα και από την ε, Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά αν δει κανείς και την ιστορία της τελευταίας πεντηκονταετίας ε, και θα δείτε τα θέματα γύρω από την αναγνώριση. Οι Τουρκοκύπροι είχαν ε, νομίζω ε, δεν, δεν ακούστηκαν ακριβώς και υπήρξαν και οι υποσχέσεις για τερματισμό της απομόνωσης του βόρειου τμήματος που δεν έχουν υλοποιηθεί. Νομίζω ότι ε, εντάξει μπορεί να υπάρχει μια μικρή μονομέρεια γιατί ζητείται από την ε, τουρκική κυβέρνηση να υποστηρίξει τι συνεχιζόμενε διαπραγματεύσει και νομίζω ότι πρέπει να πει η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση πρέπει να είναι πιο θετικέ και να υποστηρίξουν τι διαπραγματεύσει. Αλλά νομίζω ότι η παράγραφό σα είναι λογική. Κάποιες όμως από τις προτινόμενες ε, τροπολογίες δεν είναι. Το μόνο σημείο που θέλω να αναφέρω, υπάρχουν και άλλα βέβαια, αλλά το μόνο που θέλω να αναφέρω σε αυτή τη φάση, κύριε Πρόεδρε, αφορά τον ενεργειακό χάρτη. Και πάλι νομίζω ότι η παράγραφος της ΡΙΑ είναι πάρα πολύ λογική και νομίζω ότι θα είμαστε ιδιαίτερο κοντόθωροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν δεν ενθαρρύναμε το άνοιγμα του ενεργειακού ε, κεφαλαίου ε, στην περίπτωση σε αυτή τη χρονική στιγμή που όλοι προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πρόσβασή μας σε πόρους ενέργειας, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και αναγνωρίζοντας και την πολύ σημαντική θέση που θα έχει η Τουρκία σε όλη αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μεσόγειο, ε, και όλες οι προσπάθειες ε, για την εξέβρεση πετρελαιοκή θα πρέπει να γίνουν με τον λογικό τρόπο. Το να μπλοκάρει το κεφάλι για την ενέργεια νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πάρα πολύ προσοχή και να το αποφύγουμε. Χατζηγεωργίου, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι εμείς υποστηρίζουμε εν θερμά και το εννοούμε την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού πληρεί βεβαίως τα κριτήρια που έχει πληρώσει κάθε άλλο κράτος που έχει ενταχθεί. Είμαστε από εκείνου που αναγνωρίζουμε ότι πρώτα απ' όλα έχουμε συμφέρον από ένα εκδημοκρατισμό της Τουρκίας, και αυτό είναι ένας από τους κύριους λόγους που υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία τελικής ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ζητήματα όμως τα οποία πρέπει να εγείρονται γιατί κατά την άποψή μου θα είναι υποβοηθητικά για την ίδια την Τουρκία και όχι για να ασκούμε απλώς πίεση ή να τις κάνουμε κριτική. Καλούμε την Τουρκία και νομίζω αυτό είναι σωστό να απελευθερώσει τους 1.700 Κούρδους, πολιτικούς, δικηγόρους και δημάρχους που κρατούνται στις ε, φυλακές. Η ομαλοποίηση των σχέσεων της Τουρκίας με γειτονικέ χώρες, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμονίων. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι αυτή η συγκεκριμένη συγκυρία δείχνει ότι ε, καταφεύγουμε σε μια πίεση στην Τουρκία όταν συζητάμε σήμερα για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Είναι θέμα ιστορίας και η ιστορία πρέπει να αναγνωρίζεται και να διαβάζεται σωστά δεν μπορεί να διεκδικεί ρόλο ρυθμιστή στην περιοχή και να θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν συνεχίζει να παραβιάζει με στρατιωτική κατοχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το διεθνές δίκαιο και εφημεριώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελέγχθηκε εδώ ότι καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι shadow γιατί είναι παθιασμένοι οι Έλληνες ή ε, Κύπροι Ευρωβουλευτές μακάρι το εύχομαι αυτό να ήταν λιγότερο παθιασμένοι ήδη εάν τυχόν συνέβαινε στην ίδια τους τη χώρα αυτό που συμβαίνει στη χώρα την δικιά μας. Και θεωρώ ότι πολλές από τις τροπολογίες τους δείχνουν ένα ελαφρώς περισσότερο πάθος από αυτό που καταλογίζουν σε μας. Εμείς είμαστε λογικοί στις διαπραγματεύσεις και αυτό νομίζω έχει αναγνωριστεί από, από πάρα πολλούς και από την ίδια την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό πρέπει να πάψει να λέει ότι είναι υπέρ της λύσης, πρέπει να το κάνει πράξη και να ξεκολλήσει από το 2004. Οποτεδήποτε συζητήσεις με Τούρκους αξιωματούχους για τη λύση του Κυπριακού σου λέει το 4 κάναμε αυτό. Λοιπόν είμαστε στο 2011. Πρέπει να σέβεται το δίκαιο της θάλασσας. Είναι η μόνη χώρα, συνάδελφοι, στον κόσμο που δεν υπόγραψε τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Η, η μόνη χώρα. Και αμφισβητεί το δικαίωμα ενός κράτους μέλους να ενεργήσει στην δική του οικονομική ζώνη έρευνες για έβρεση υδρογοναθράκων. Το θέμα της Αμοχώστου είναι μια πόλη η οποία κάθεται εκεί 36 χρόνια. Πρέπει να υπάρξει απέτηση να επιστραφεί η πόλη στους κατοίκους. Και για το θέμα των αγνοωμένων θέλω να πω μια φράση. Υπάρχει εξέλιξη αλλά πρέπει να πιεστεί η Τουρκία να δώσει πληροφορίες από τα αρχεία της ε, του 1974 για να βρούμε την τύχη όλων των αγνοωμένων της Κύπρου. Ευχαριστώ. Ε, ε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συγγήτρια θέλει να είναι ισόρροπη η έκθεση και ζητά κάποιες τροπολογίες να αποσυρθούν. Ακούγοντας όμως ε, τις άλλες ομάδες και τη διάθεση δεν με προδιαθέτει αυτό να αποσύρω τροπολογίε, γιατί θεωρώ ότι είναι καθήκον μα, όχι μόνο δικαίωμά μα, αλλά και καθήκον μα ω Κοινοβούλιο να ασκήσουμε και να παρακολουθούμε επικριτικά τι εξελίξει στην Τουρκία. Και νομίζω ότι ένα σημαντικό τομέα όπου διαπιστώνουμε ότι δυστυχώ έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα από τότε που ξεκίνησε η Τουρκία το 2005 τι διαπραγματεύσει. Και να σα πω και το έκθεση προόδου θεωρώ αποτελεί εφημισμό. Ονομάζουμε κάθε φορά έκθεση πρόοδου την έκθεση αυτή. Θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα να ανα, αναφέρω ότι η 395, η 295, η τροπολογία για την τροπολογία 39, για την ε, έκθεση 39 της ε, έκθεσης για την στάση της Τουρκίας ως προς το Ιράν και τα πρινικά όπλα θα ήθελα να, να αποσύρω Και εγώ λυπάμαι που ψήφισε κατά η Τουρκία του σχετικού ε, ψηφίσματος του ΟΗΕ. Θα ήθελα λοιπόν να την αποσύρω την τροπολογία αυτή, να είναι μόνο του κυρίου Μάλτσερ πλέον αυτή η τροπολογία. Ευχαριστούμε κύριε Κλάσα. Θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους ε, συναδέλφους που έχουν ζητήσει το χρόνο, γιατί θα πρέπει να μειώσω σε ένα λεπτό τον χρόνο αγόρευσης είναι πολύ εγγεγραμμένη. Κύριε Κόβατσεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Ουμεν για την καλή δουλειά που έχει κάνει ε, μέχρι τώρα είναι ε, γεγονός ότι θέλουμε μια Τουρκία η οποία θα έχει κάνει ανακοχή, θα έχει συμφιλειωθεί με τις ε, ε, γείτονες χώρες και η οποία θα δουλέψει προς τη δημοκρατία, προς τις καλές σχέσεις, φιλικές σχέσεις με τους, με τους γείτονες, προς τη δημοκρατία και προς τα σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να εργαστεί λοιπόν και να εργαστούμε και εμείς στενά σε συνεργή συνεργασία με την ε, Τουρκία ε, έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να λύσουμε και το πρόβλημα της Κύπρου αλλά και το πρωτόκολλο της Αρμενίας και με συμφωνώ με την Ρίτα με όλα αυτά που είπε προηγουμένως και βεβαίως ε, νομίζω ότι ε, δεν είναι δυνατόν να μην ξεχνάμε και τις ε, προσπάθειες συμφιλίωσης που έχουν γίνει και από την πλευρά του κυρίου Ερντογάν όσον αφορά το θέμα της της Αρμενίας. Επίσης υπάρχει η συνθήκη της Αγγόλας και έχουμε και άλλα πιο πρόσφατα νέα. Η συμφωνία επανεισδοχής έχει ήδη ε, βρεθεί σε τελική φάση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και Τουρκίας. Ε, υπάρχουν οι συμφωνίες για τον αγωγό Ναμπούκο και νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να μπουν στην διαδικασία συμφιλίωσης και να μην παραμείνουμε προσκολλημένοι σε προβλήματα του παρελθόντος. Κυρία Κοπά, παρακαλώ ένα λεπτό. Μικρόφωνο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια και να αναγνωρίσω τη δύσκολη δουλειά που την περιμένει με τόσες τροπολογίες. Νομίζω σημασία έχει το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές πως δεν επιθυμούμε τα διέξοδο στην ενταξιακή πορεία και να επιβεβαιώσουμε τις δεσμεύσεις που απορρέουν για το διαπραγματευτικό πλαίσιο τόσο για την ευρωπαϊκή πλευρά όσο για την Τουρκία πρέπει να είμαστε έντιμοι και να αναγνωρίσουμε τα σημεία όπου υπήρξε πρόοδο, όπως το θετικό βήμα τη συνταγματική αναθεώρησης όπως και οι συμβολικές ε, σημασίες εξελίξει εξελίξεις στο ζήτημα των θρησκευτικών ελευθεριών. υπάρχουν όμως σημεία όπου δεν σημειώθηκε καμία πρόοδο και το κυπριακό είναι το πιο κλασικό παράδειγμα και εκεί νομίζω το πιο σόφρον είναι να παραμείνουμε στι περσινέ διατυπώσει. Ε, παρά τις προσπάθειες τέλος για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι γεγονός ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της χώρας μου παραμένουν καθημερινό σχεδόν φαινόμενο. φανταστείτε να ζείτε σε ένα μικρό νησί και κάθε μέρα μαχητικά αεροσκάφη να πετούν σε χαμηλό ύψος πάνω από τα σπίτια. θέλω λοιπόν να τονιστεί στη φετινή μας έκθεση ότι παρόμοιες πράξεις δεν συμβιβάζονται ούτε με διακηρυγμένη πολιτική μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες του κ. νταβούτογλου ούτε με την υποχρέωση καλής γειτονίας με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κάζακ, ένα, λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ρόιτεν για την έκθεσή της το ότι υπάρχουν τόσες ε, τροπολογίες ε, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο περίεργο ε, δεδομένων και των εκθέσεων που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Έχω καταθέσει και εγώ κάποιες τροπολογίες και μάλιστα συγκεκριμένα πρότεινα στις αιτιολογικές σκέψεις να αναφέρεται η έγκριση από το Κοινοβούλιο μιας έκθεσης για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία αναφέροντας ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις ε, διαβατηρίων, είναι ένα μείζον ζήτημα, όπως γνωρίζετε. Όταν υπάρξει πια η Συμφωνία Επανεισδοχή, νομίζω θα είναι πια καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει αίσθημα υπευθυνότητα και να, να απλουστεύσει για τους επαγγελματίες, για τους φοιτητές τουλάχιστον ε, το καθεστώς χορήγησης ε, θεώρησης διαβατηρίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, νομίζω ότι επίση είναι καιρό πια να γίνει μια ειλικρινή και μεγάλη ανοιχτή συζήτηση για όλο αυτό το ε, πολύπλευρο ζήτημα του Κυπριακού. Πρέπει να θυμηθούμε ότι δεσμεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 για να τεθεί ένα τέρμα στην απομόνωση τη τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τάνοκ, για ένα λεπτό θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια για την ισορροπημένη έκθεση ένα τόσο ε, λεπτό ζήτημα της ε, πολιτικής. Εμένα με αφορά ε, το θέμα κάποιων θρησκευτικών μειονοτήτων όπως είναι η Ασσύριοι, παραδείγματος χάρη και το τι πρέπει να γίνει και παρά τις υποσχέσεις δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα από την τουρκική ε, κυβέρνηση. Και επίσης ε, υπάρχουν ε, και πολλές εξηγήσεις που πρέπει να δώσει για το γεγονός ε, των εορτασμών ή μη εορτασμών του τουρκοκυπριακού εδάφους που ε, δηλαδή απαγόρευσε να εορταστεί ε, τα Χριστούγεννα. Θα δούμε τι θα προκύψει και με την επίσημη έκθεση. Ξέρουμε ότι μπλοκάρει επίσης ε, και τη συνεργασία με τον άτομο στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ και έχουμε και τα πρωτόκολλα αυτά τα οποία δεν τηρούνται. Έχουμε την εχθρότητα απέναντι στην κυβέρνηση της Κύπρου και ο κύριος Έρογλου ουσιαστικά δείχνει να μην θέλει να υπάρξει μια ρύθμιση η Τουρκία ε, ούτε για την αμόχωστο κάνει μία κίνηση καλής θέλησης όπως θα έπρεπε να κάνει για την ε, ε, για τις διαπραγματεύσεις. Παραμένουν ε, τα θέματα αυτά ανοιχτά και σε ό,τι αφορά την Αρμενία δεν ε, αναγνωρίστηκε η γενοκτονία των Αρμενίων. Εγώ θέλω να υποστηρίξω τις τροπολογίες ε, που κάνουν τη σχετική αναφορά και πρέπει να δούμε και τι γίνεται και με τον Αγκόρνο Καραμπάχ που είχε πει του και πέρυσι ότι υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας. Πρέντα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ την εισηγήτρια για τον τρόπο με τον οποίο συνέταξε την έκθεσή της. Έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες και θα ήθελα να εξηγήσω το πνεύμα των τροπολογιών αυτών. Όσον αφορά το άρθρο 2 ε, για το οποίο ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις, λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν πλέον, να ανοίξει το κεφάλαιο, έτσι ώστε να έχουμε πραγματική συζήτηση έτσι ώστε η Τουρκία να μπορέσει να μεταφέρει ε, το κοινοτικό κεκτημένο. Επίσης ε, θα ήθελα να σημειώσω την πρόοδο ε, της Τουρκίας όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, όσον αφορά κάποια τεχνικά στοιχεία. Ομοίως να υπογραμμίσω ότι το κεφάλαιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαιοσύνη πρέπει να ανοίξει έτσι ώστε να έχει κίνητρο η Τουρκία να προοδεύσει όσον αφορά τα θέματα αυτά. Επίσης πρέπει να χαιρετήσουμε την στήριξη της Τουρκίας όσον αφορά ε, την ε, αντιπυραυλική ασπίδα. Ευχαριστούμε πολύ ε, κύριε Πρέντα γιατί είσαστε ο μόνος που δεν ξεπέρασε το χρόνο σας Πάτσκουρ. Κυρία Μποσκούρτη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τη Ρία, να ευχαριστήσω για τις ε, ιδιότητες που μου ε, αποδίδεις ε, σε ό,τι αφορά μια διμερή ε, συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ωστόσο χαίρομαι με τη συμφωνία για την επανεισδοχή ε, λαθρομεταναστών. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνοδευτεί και με μια ε, γρήγορη εκκίνηση των συζητήσεων για τις θεωρήσεις με, τις, με την Τουρκία σε ό,τι αφορά το πόσο φιλόδοξοι θα πρέπει να είμαστε. Συμφωνώ με τη Ρία ότι θα πρέπει να δείξουμε ένα όραμα για το μέλλον. Ε, βλέπω ότι βασικά ε, υπάρχει μια συσσόρευση παλαιού πόνου, αν θέλετε. Θα πρέπει όμως να κοιτάξουμε και προς το μέλλον, να στραφούμε και προς το μέλλον. Νομίζω ότι ως κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Να δούμε ως κοινοβούλιο πως μπορούμε να προχωρήσουμε με την Τουρκία και πως μπορούμε να προχωρήσουμε γενικότερα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με επικοδομητική ε, στάση. Κατσίν για ένα λεπτό. Ο κύριος Κατσίν δεν είναι εδώ και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντάφ για ένα λεπτό. Um, uh, Ευχαριστώ και συγγνώμη. Λυπάμαι. Νομίζω ότι ήταν μοιραίος ο συνδυασμός τριών παραγόντων, ο οποίος ουσιαστικά βήθησε ή τουλάχιστον ε, καθυστέρησε τη διαδικασία προσχώρηση. Καταρχάς, η φτωχή απόδοση, επίδοση του Συμβουλίου. Κατά δεύτερον, η συνεχιζόμενη ε, ιδεολογία του κεμαλισμού στην Τουρκία. Και τρίτον, η στάση και των δύο πλευρών που είναι ατυχής και ε, για, την Κύπρο. Νομίζω ότι αυτά τα τρία στοιχεία συντελούν στο να μην μπορεί να γίνει φέτος μια χειρονομία ουσίας και από τις δύο πλευρές. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η διαδικασία προσχώρησης έχει βυθιστεί και ότι την ίδια εποχή του χρόνου θα αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε εναλλακτικά, μια εναλλακτική λύση ως προς την ε, ε προσχώρηση. Ευχαριστώ κύριε Ντάφ. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Ένα λεπτό επίσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την εργασία ποιότητα που έκανε η κυρία Ρούιτεν. Κατανοώ τον προβληματισμό τη για το μεγάλο αριθμό των τροπολογιών, αλλά ταυτόχρονα είμαι σίγουρο ότι θα φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα αποδεκτό από τη μεγίστη πλειοψηφία των συναδέλφων. Ορισμένε επισημάνσει θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι με την Τουρκία, αναφίβολα. Αυτή είναι η προπόθεση για να μπορούμε να είμαστε και αυστηροί στα σημεία που οφείλουμε να είμαστε αυστηροί εξαιτία καθυστερήσεων, αδυναμιών, τη επιφυλακτικότητα και πολλέ φορέ τη άρνηση τη Άγκυρα να ανταποκριθεί στα κριτήρια και τα προαπαιτούμενα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από αυτά είναι η υποχρέωση τη Τουρκία να υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο τη θάλασσα. Η σύμβαση αυτή, κύριε Πρόεδρε, αποτελεί κοινοτικό κεκτημένο η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλόμενο μέρος στη σύμβαση αυτή. Όλα τα κράτη-μέλη και τα 27 την έχουν επικυρώσει, καθώς και όλα τα υποψήφια κράτη-μέλη, με μία εξαίρεση, την Τουρκία. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει χωρίς άλλη καθυστέρηση τη σύμβαση αυτή. Το άλλο θέμα είναι οι σχέσεις καλής γειτονίας. Σε αυτό είναι απαραίτητο να σταματήσει η σταθερή και επικίνδυνη πρακτική της παραβίασης εθνικού εναέριου χώρου ενός κράτους μέλους της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουμουτσάκο. Ο κύριος Μαυρονικόλας, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω την ευαρέσκεια μου για το ισορροπημένο κείμενο της εισηγήτριας και παράλληλα για τον ισορροπημένο τρόπο που αντιμετωπίζει πολλά από τα θέματα τα οποία αφορούν την Τουρκία. Θα ήθελα από τη δική μου πλευρά μέσα στις πραγματικότητες του κυπριακού προβλήματος να ζητήσω να γίνει αντιληπτόν ότι ορισμένες προσθήκε οι οποίες αφορούν κυρίως την προσπάθεια επικοινισμού των κατεχομένων όπως επίσης ορισμένες προσθήκες που έχουν σχέση με το να δοθεί η αμόχωστος πίσω στους κατοίκους της αποτελούν αδιάσυστα στοιχεία του κυπριακού προβλήματος και αναφίβολα και της απόφασης που θα έχουμε σε σχέση με την Τουρκία. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το κεφάλαιο της ενέργειας μπορεί να ανοίξει μόνον τότε όταν η Τουρκία αρχίσει να σέβεται γειτονικά κράτη, να σταματήσει να παρενοχλεί κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα και η Κύπρος στις ανάλογες έρευνες τις οποίες κάνουν. Και παράλληλα θα ήθελα τελειώνοντας να αναφέρω ότι οι εισηγήσει ιδιαίτερα από την κυρία Φλότρου των Πρασίνων που εμπεριέχουν ξανά το σημείο του απευθείας εμπορίου με τα κατεχόμενα που περιέχουν την ονομασία της Βορείου Κύπρου με υπονοούμενο αναγνώριση, είναι έξω από τις πραγματικότητες του σημερινού κυπριακού προβλήματος και των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Παπαδοπούλου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εμπιστεύομαι ότι η κυρία Όμεν θα καταφέρει να βρει συνενετικέ διεξόδου στι προτενόμενε 315 τροπολογίε. Προσωπικά αποσύρω την τροπολογία 215 για την Αρμενία, υποστηρίζοντα τι τροπολογίε 220 και 218. Δεν μπορώ να αποσύρω τροπολογίε για την Κύπρο όμω, γιατί εδώ έχω δει αρκετέ τροπολογίε που δυστυχώ προσπαθούν να παραγράψουν παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια προσπάθεια απενοχοποίηση τη Τουρκία βουλευτέ θέλουμε να καταγράφονται πραγματικά γεγονότα και τα γεγονότα στην κύπρο μιλούν ότι η τουρκία παραβιάζει γιατί προχωρεί σε παράνομον επικισμών, θυματοποιεί ελληνοκύπριου και τουρκοκύπριου δεν έχει υλοποιήσει το πρωτόκολλο και αυτέ είναι ευρωπαϊκέ υποχρεώσει οι οποίε στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται. επίση η παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών σε βάρο των ελληνοκυπρίων δυστυχώ έχουν αυτόν παράδειγμα γιατί τα χριστούγεννα τερματίστηκε η χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο κατεχόμενο ριζοκάρπασο. Αυτά πρέπει να καταγραφτούν στην έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαδοπούλου. Έχουμε ακόμα πέντε λεπτά έτσι ώστε η συγγήτρια, ε, η κυρία Όουμεν Ρόιτεν, να απαντήσει. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Να πω προς τους συναδέλφους Καταρχάς ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία αυτή που θα πρέπει να έχει δίκαιη και επικριτική αντιμετώπιση, αλλά αυτό θα προσπαθώ να το κάνω και προς τους συναδέλφους, να είμαι επικριτική και δίκαιη. Μία παρατηρήση ακόμα να κάνω, Πρόεδρε. Το 2006, όχι, όχι, είναι η τέταρτη έκθεση. Στην πρώτη έκθεση μου ξεκίνησα κάνοντας κάποιες ε, παρατηρήσεις για διμερή ε, ζητήματα μεταξύ Τουρκίας και, άλλων χωρών. Εκτιμήθηκαν αυτές οι παρατηρήσεις και κάθε χρόνο κάνω κάτι διαφορετικό. Αλλά πάντα σε όλες τις παρατηρήσεις επανερχόμαστε. Να σας ε, προειδοποιήσω και να πω στους συναδέλφους ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί απαραίτητα αυτή τη φορά. Δεν θα επαναλάβουμε αυτά που είπαμε τις προηγούμενες χρονιές. Πρόεδρε, ό,τι μπορεί να συνδράμει στην επίλυση, του προβλήματα, στην επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στην ε, νήσο, θα τα κάνω. Αλλά δεν έχει νόημα να διευρύνουμε τις διμερείς διαμάχες. Κατά δεύτερον, σε... για τις παρατηρήσεις ε, για την ε, προσχώρηση, θα είμαι δίκαιη, τίμια και θα αντιμετωπίσω τα πράγματα με συνοχή. Και για τον συνάδελφο Μπρέιντα, γιατί αναφέρθηκε σε κάποιες τροπολογίες ως προς τον ανταγωνισμό. Στον ανταγωνισμό. Πρόκειται για το κεφάλαιο που αντιμετωπίζει η... Συγγνώμη, πρόκειται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η οποία δεν είναι έτοιμη, μπερδεύτηκε η ομιλήτρια και ανέφερε την Ελλάδα. Ζητάμε να ανοίξουν κεφάλαια όπου δεν είναι τεχνικά δυνατόν αυτό. Στην ε, ατμόσφαιρα αυτή να θα είμαι ανοιχτή και επικριτική Ελάτε συνάδελφοι, θα σας υποδοχτώ με μια κούπα καφέ και θα σας αποδείξω ότι είναι καλύτερο να κοιτάξουμε το μέλλον σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Ούμεν ε, Ρόιτεν. Μας ε, βοηθήσατε έτσι ώστε, γιατί δεν μιλήσατε πολύ, ε, να σας πω ότι η ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή στις 10 Φεβρουαρίου και θα περάσει στην Ολομέλεια τον μήνα Μάρτιο. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ μια και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σας παρακαλώ λέγω να βάλετε την ε, ε, καρτέλα σας στο μηχάνημα. Έχουμε την ε, ψηφοφορία της έκθεσης Μπέλτερ προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Ιράν. Έχουν υποβληθεί 301 τροπολογίες, έστω και αν υπάρχουν πολλές ταυτόσιμες. Επίσης, μέσα από, συμβι... μέσα από συζητήσεις και συναντήσεις, ο εισηγητής έχει υποβάλει 18 συμβιβαστικές τροπολογίες και είναι υπέρ των περισσότερων. Μπορούμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ξεκινούμε με τον ε, συμβιβασμό 4. Συμβιβασμός 4. Ψήφι υπέρ. Υπέρ. Υπέρ. Συμβιβασμός 4. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μου λένε ότι από τη στιγμή που η 78 απερίφθη ε, έπρεπε να ψηφίσουμε και τις ενδιάμεσες τροπολογίες. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 79 και 80 ως ταυτόσημες υπέρ. 79 και 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για... Θέλετε να γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία για το 84. Ωραία. 84 διελεκτρονικής ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. θέλε 84 ηλεκτρονική ψηφοφορία για να ελέγξουμε το αποτέλεσμα πέρα της ψηφοφορίας 32 κατά 24 υπέρ και νομίζω ότι έχουμε ακόμα μία ε, ψήφο κατά, ναι, 24-33 ε, κατά, ε, απορρίπτεται. Η 85 έχει αποσυρθεί, 86 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 87, 88, 89 ταυτόσιμε τροπολογίε. ψηφίζουμε υπέρ, κατά. αποχέ εγκρίνονται 91 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τις ψηφοφορίες, λείπει μία ψήφος, δεν πειράζει. 26 κατά 34 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογίες 90, 92, 93 ψηφίζονται από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103, 104, 105 και 106 από κοινού υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 107 Θέλετε έλεγχο ηλεκτρονικό, πολύ ωραία. 103, 104, 105, 106, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. 31 ψήφοι κατά, 34 ε, υπέρ, εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στο συμβιβασμό 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108. Τροπολογία 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. έχουμε μία προφορική τροπολογία. Είναι γραμμένο στο κατάλογο ψηφοφορίας μας, άρα δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109-115 υπέρ. Ο κύριος Σάκ θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Σάκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι δύσκολο το θέμα, γιατί βεβαίως όλοι καταδικάζουν ε, την, τον απαγχωνισμό της ε, Ιρανής ε, με Ολλανδική υπηκότητα της κυρίας Σαράνη αλλά ε, το θέμα δεν είναι μόνο η δική της περίπτωση. Εμάς μας ενδιαφέρει ε, οποιαδήποτε θανατική καταδίκη ε, είχαμε πει ότι δεν θα αναφέρουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή την αρχή. Όχι επειδή θεωρώ ότι η περίπτωση της κυρίας Μπαχράμη δεν είναι ε, ε, τρομακτική. Λαμβάνουμε υπόψη, ναι, λέει ο Πρόεδρος, όχι, όχι, προσπάθησα από πριν να κινήσω την προσοχή σας. Ήθελα να μιλήσω πριν από την ψηφοφορία για να πω ότι δεν θα ήθελα να γίνει δεκτή αυτή η ε, ψηφοφορία. Ναι, ε, κοιτάξτε λέει ο Πρόεδρος, δεν μπορώ να ξεκινήσω συζήτηση πάνω σε αυτό. Ε, λυπάμαι εάν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα θέλατε εσείς, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Ψηφίζουμε την 109-115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ α, ηλεκτρονική επαλήθευση 109-115 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας 37 ψήφοι κατά συν 1 38, 29 υπέρ, επομένω απορρίπτεται, 114 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται, 119 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 120, 121, 122 ταυτόσημες ψηφίζονται από κοινού υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνονται. 126, 127, 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140-141 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147-212 από κοινού γιατί ταυτόσιμε ταυτόσιμες τροπολογίες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 149-150-151 είναι ταυτόσιμες ψηφίζονται από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 έχει αποσυρθεί, συμβιβασμός 9 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται, 160 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 161, 162, 163 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται 164 Λοιπόν, ωραία, η ηλεκτρονική επαλήθευση για τις τροπολογίες 161, 162, 162 που ψηφίζονται από κοινού. Η Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, είναι θετική η έκβαση. 35 υπέρ 33 ψήφοι κατά, επομένως ε, εγκρίνονται. 166, 167, 168 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 172, 173, 174 ταυτόσιμες από κοινού υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. 175 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. 176 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 183 μαζί με το 184-185 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 Υπάρχει εδώ προφορική τροπολογία η οποία σας έχει μοιραστεί. Δεν ξέρω εάν κάποιος συντονιστής... Κύριε Γκάλερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο σκοπός είναι, αν συμφωνήσουμε, να αποσύρουμε την 188 και θα ήθελα στη μέση να μπουν, να μπει η διατύπωση προκειμένου να βάλουμε έναν όρο σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις με την κοινωνία των πολιτών. Αυτός είναι ο όρος και μετά την τελεία να καταστεί αυτό προαιρετικό και να ζητήσουμε και συναντήσεις με πολιτικούς κρατήμενους. Αυτό όμως δεν θα είναι όρος. Άρα να αναφέρουμε, τονίζει ότι οι επισκέψεις των ε, εκπροσώπων των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποτελούν ε, υπό τον όρο μάλλον με τι συναντήσει με εκπροσώπου τη κοινωνική των πολιτών και ότι θέλουμε να υπάρχουν και επισκέψει με κρατούμενου. ιδιαίτερα αυτού που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο. Μόνο και Βανόρντεν έχουν ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με το άρθρο 156.6 του κανονισμού Είμαστε αντίθετοι στην υποβολή προφορικής τροπολογίας όταν πλέον ε, έχουν συμφωνηθεί συμβιβασμοί και έχουμε επεξεργαστεί προηγουμένως προφορικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Φαν συμφωνώ, συμφωνώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τις επισκέψεις αυτές. Υπάρχει ένα λόμπι, για τις βίζες, συγγνώμη. Υπάρχει ένα λόμπι που προσπαθεί να ε, χρησιμοποιήσει αυτό το θέμα. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι προπαγάνδας για τους οποίους χορηγούνται ε, αυτές τις θεωρήσεις και νομίζω ότι η προφορική αυτή τροπολογία, επισκέψεις μάλλον, ε, πρέπει να μην γίνει δεκτή. Ναι, δεν μπορούμε να ανοίξουμε όμω την ε, συζήτηση γιατί ε, η παρέμβαση τη κυρία Μούνη που είναι διαδικαστική απαγορεύει οποιαδήποτε συζήτηση. Επομένω, θα ψηφίσουμε την τροπολογία ω έχει. Είναι διαδικαστικό το ζήτημα. Δεν μπορώ παρά να το σεβαστώ. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 187 χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ κατά, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, ηλεκτρονική επαλήθευση. 187 άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εάν θέλετε να κοινοποιήσετε την θέση της ομάδας, κύριε Γκάλερ, ε, παρακαλώ μπορείτε να το κάνετε. Εάν θέλετε, λέω, να μας πείτε ε, την θέση της ομάδας, γιατί, δεν, γιατί ψηφίζουμε την τροπολογία χωρίς τη δική σας προφορική τροπολογία. Η εντύπωσή μου από πλευρά της ομάδας μου είναι ότι χωρίς την ε, προφορική τροπολογία δεν υποστηρίζουμε πλέον την τροπολογία. Αυτά. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η, η ψηφοφορία και απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 188. Ψηφίζουμε 188 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται 190 Α, η ηλεκτρονική επαλήθευση 189 η ηλεκτρονική επαλήθευση για το 189 πέρας εγκρίνεται 37 ψήφοι υπέρ 32 κατά 190 Όχι, όχι. Πηγαίνουμε στο συμβασμό 11 από τη στιγμή που ε, είχαμε ψηφίσει το 189. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 200 201 ταυτόσημες υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 203 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 202-204 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 213 πρέπει να δώσουμε τον λόγο σε όποιον θέλει από το ΕΛΚ να αναφερθεί στην προφορική τροπολογία. Στη γραμμή που ζητήσαμε και προηγουμένω θέλουμε να, να διαγράψουμε την τελευταία πρόταση επειδή αναφέρεται σε μεμονωμένε περιπτώσει, Προτείνουμε λοιπόν να διαγραφεί η τελευταία πρόταση, η τελευταία φράση. Η κυρία Ράιτον, ευχαριστώ. Ναι, εγώ υπέβαλα την τροπολογία. If, if anybody, if anybody... Αν είχε έρθει κανείς σε επαφή μαζί μου, θα είχε λάβει την απάντηση που θα σας δώσω τώρα, ότι είναι απαράδεκτο γιατί η κυρία αυτή εκτελέστηκε διαπαγχωνισμού την Κυριακή. Γιατί να μην ζητήσουμε από την υπότιτλη εκπρόσωπο κάτι να κάνει για την τεράστια αυτή απειλή. Διαφωνώ. Και θέλω να ψηφιστεί. <laughs> Ναι, και σε αυτή την περίπτωση, όπως γνωρίζετε, συνάδελφοι, ησυχία. Και σε αυτή την περίπτωση, μονάχα ένα συνάδελφος να πει ότι είναι κατά έτσι ώστε να μην ε, συμπεριληφθεί η προφορική τροπολογία. 213 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 218 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ψηφίζουμε 218 ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 218 218 ηλεκτρονική ψηφοφορία λείπουν τρεις συνάδελφοι κλείνουμε την ψηφοφορία 36 υπέρ, 32 κατά, επομένως εγκρίνεται. Ε, Συμβιβασμό 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 229 κατά τμήματα υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα 229 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 14 υπέρ Α, θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 229. Δεύτερο τμήμα, λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τριάντα υπέρ, 40 κατά απορρίπτεται. Συμβιβασμός 14. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 234-35-36 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Άρχεται η ηλεκτρονική επαλήθευση επί των τροπολογιών 35 236 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 34 ε, κατά, 36 υπέρ, επομένως εγκρίνεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 238 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 239, 240 συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ. Κατά Ούτε εδώ είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση 241. Άρχεται η ψηφοφορία. Τρεις συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Τώρα ένας <laughs> έμεινε, τώρα ψήφισαν όλοι. Πάρα πολύ ωραία. 36 υπέρ, 33 κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 258 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 259 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 261 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 213 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 264 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 265 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 17 Α, 265 θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Άλλη φορά δεν θα χρησιμοποιώ ε, την... Ε, θα χρησιμοποιώ την οριστική έγκληση μονάχα. Εγκρίνεται, όχι μάλλον εγκρίνεται. Πέρα στις ψηφοφορίες, 37 ψήφοι κατά, 33 υπέρ, άρα δίκιο είχα που είπα μάλλον. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 281 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μα, απορρίπτεται διορθώνει Πρόεδρος. 282 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 283 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 284 έχουμε και εδώ προφορική τροπολογία Λαντσμπέργκης έχει το λόγο. Εσείς κύριε Λαντσμπέργκης έχετε το λόγο. Κύριε... κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να προτείνω μία απλουστευμένη εκδοχή. Μετά από εκεί που λέει συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων, να λέει κατά καταβλισμών Ιρανών προσφύγων κτλ. Κυρία Μούνιθ, είμαστε κατά της προφορικής τροπολογίας, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα και προηγουμένως, αρκεί ένας συνάδελφος να αντιτίθεται στην προφορική τροπολογία, ε, ε, ώστε να μην έχουμε τη δυνατότητα να το συμπεριλάβουμε. Άρα ψηφίζουμε τη 284 ως έχει, χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 287. 6. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 287. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 295. Μαζί με τη 296 και 297 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αμφιβάλλω για το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 295, 296 και 297 που είναι τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες. Πέρας της ψηφοφορίας, 33 ψήφοι κατά, 35 ψήφοι υπέρ, άρα εγκρίνεται 299 υπέρ Λίγοι μου φαίνονται αυτοί που είναι υπέρ. Κατά, αποχές, σαφώς απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2. Είναι γραμμένο στον ε, κατάλογο ψηφοφορίας υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 301 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 22. Δύο δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Αφαιρέθηκαν μάλλον. Τροπολογία 22. Αλλά ας κλείσουμε. Κλείνουμε λοιπόν την ψηφοφορία. 34 ψήφοι υπέρ, 35 κατά. Απορρίπτεται. «23 υπέρ» «κατά αποχές απορρίπτεται». 24 ε, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 έχει αποσυρθεί, 32. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Εντάξει, επί της 30. Και εγώ δεν ήμουν σίγουρος. 30, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 30. Τώρα ψήφισαν όλοι. Πέρας. 35 κατά, 34 υπέρ, άρα απορρίπτεται με διαφορά μιας ψήφου. Απορρίπτεται. Έχει αποσυρθεί η τροπολογία 31. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 32. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 32 πέρας 35 υπέρ 34 κατά αυτή τη φορά εγκρίνεται με διαφορά μίας ψήφου δεν ψηφίζουμε 33 η 35 έχει αποσυρθεί επομένως 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 απεσύρθη 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος ηλεκτρονική Ψηφοφορία επί της τροπολογίας 42, ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας της ψηφοφορίας. 29 κατά 40 υπέρ εγκρίνεται. 43 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογίες 54-55 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος ωραία επαλήθευση για την τροπολογία 57 άρχεται η ψηφοφορία «29 ψηφίσαντες, 34 υπέρ, 35 κατά για μία ψήφο απορρίπτεται. 58 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64-65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 Α, ε, θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση 64-65 64-65. Υπάρχει ένας συνάδελφος που δεν έχει ψηφίσει, αλλά παρόλα αυτά κλείνουμε την ε, ψηφοφορία. 31 ψήφοι υπέρ, 33 κατά απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται νομίζω. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 5. Η 3 απερίφθη και επομένως πρέπει να ψηφίσουμε και την τροπολογία 4. Άρα ψηφίζουμε πρώτα την 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 5 παρακαλώ πολύ. Πέρας. 32 ψήφοι υπέρ, 37 κατά, επομένως απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Έχει αποσυρθεί η 7. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 10-11 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω. Συμβιβασμός 1 υπέρ. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για το 10 και 11. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 10 και 11. Πέρας. 31 ψήφοι υπέρ, 34 κατά, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας 62 υπέρ, 3 ψήφοι κατά, 2 αποχές Συγχαρητήρια. Ορίστε εδώ, θριάμβευσε ο συνάδελφος Μπέλντερ πάλι. Ο κύριος Σαλαφράγκα ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ κύριε Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα απλά να πω ότι στην Επιτροπή μας ακολουθείται πάντοτε μια πρακτική, μια συμφωνία κυρίων, βάσει της οποίας πάντοτε γίνονται δεκτές ή προφορικές τροπολογίες και δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός. Λάβαμε υπόψη μας και σημειώσαμε ότι κάποια πολιτική ομάδα δεν τήρησε τελικά αυτή τη συμφωνία κυρίων. Θα κάνουμε και εμείς το ίδιο σε αντίστοιχες άλλε ψηφοφορίε. Νομίζω ότι Καλό είναι να γίνονται δεκτέ προφορικέ τροπολογίε. Οι δικέ μα προφορικέ τροπολογίε αποφασίστηκαν σήμερα το πρωί και νομίζω ότι σε καλό πνεύμα θα μπορούσαμε ε, δημοκρατικά να το κάνουμε αυτό. Αλλά αφού έτσι κατά πρόσωπο μας ε, έφεραν τον κανονισμό ως πρόσχημα, θα το κάνουμε και εμείς σε όλες τις άλλες ψηφοφορίες. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό που είπατε, έχετε δικαίωμα να πείτε αυτά που είπατε, αλλά εγώ έχω μπροστά μου μόνο τον κανονισμό. Αρκεί ένα συνάδελφο να μην είναι ε, σύμφωνο με την ε, αποδοχή μια προφορική τροπολογία και εγώ δεν μπορώ να την αποδεχτώ. Ε, ε μερικές φορές υπήρξε όντω μια συμφωνία μεταξύ των ομάδων και ίσω αυτό είναι θετικό, αλλά τη στιγμή που κάποιο δεν εφαρμόζει αυτήν την καλή α πούμε, συμφωνία, συμφωνία. Ε, δυστυχώς εγώ πρέπει να δεχτώ την κατάσταση ω έχει. Θα δώσω τώρα την Προεδρία στον κύριο Πάσκου και εγώ σας χαιρετώ. Υπόθεση.

Now <clears throat> we shall um, pass to the discussion of amendments and the report. Να περάσουμε στη συζήτηση των τροπολογιών και για μια έκθεση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το Συμβούλιο και τον κόλπο. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μποντή να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην έκθεση αυτή το μήνυμα που θελήσαμε να εκπέμψουμε είναι ότι πρέπει εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου να αναπτύξουμε και να εμβαθύνουμε τις πολιτικές μας σχέσεις. Οι τομείς πιθανής συνεργασίας είναι πολυάριθμοι και γι' αυτό Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έλθουν σε αίσιο πέραση ατέρμονες διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και 20 περίπου χρόνια για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας ελεύθερων ε, συναλλαγών. 72 τροπολογίες έχουν κατατεθεί για την έκθεσή μου και θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές οι οποίοι είχαν την ευγενή καλοσύνη να εμπλουτίσουν το κείμενο αυτό. Και όλος ιδιαίτερος θέλω να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία τους. Άλλωστε πολλές από τις τροπολογίες κατέληξαν σε μια συμβιβαστική λύση την οποία φαντάζομαι ότι θα στηρίξει η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων. Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν αφορούν κυρίως πέντε μεγάλα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, ανθρώπινα δικαιώματα. Δεύτερον, θέματα διπλωματικά, περιφερειακά, διαμεσολάβηση. Τρίτον, διαθρησκιακός διάλογος. Τέταρτον, προβολή ορατότητα της ε, δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ρόλου που μπορεί και πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τέλος ανάπτυξη διμερών σχέσεων. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολλές τροπολογίες μεταφράζουν σε χαρτί και μελάνι μια μεγάλη ανησυχία των συναδέλφων για τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα, καταπολέμηση των διακρίσεων που εν μέρη ε, έχει να κάνει με τη θρησκεία ή το ότι τα έλογα άτομα μπορεί να ανήκουν σε μια μειονότητα. Και επίσης από τις τροπολογίες αυτές αποκαλύπτεται μεγάλη ανησυχία σε σχέση με την κατάσταση των μεταναστών, των, των οικονομικών μεταναστών συγκεκριμένα. Και υπάρχει ε, και η κατάφορη αντίθεσή μας ως Ευρωκοινοβουλίου στη θανατική ποινή καθώς και στον ακροτηριασμό, τιμωρίες που δυστυχώς εξακολουθούν να ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Πρέπει παρόλα αυτά να υπογραμμίσουμε ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου εδώ και κάποια χρόνια ε, έχουν κάποιες νέες διαδικασίες ε, εισαγάγη πολιτικού και κοινωνικού εξυγχρονισμού. Αυτό συνιστά μια δυναμική την οποία νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε. Οι προσπάθειες τις οποίες, ε, τις οποίες έχουν ξεκινήσει οι χώρες του κόλπου για τα θέματα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσουν και ένα θέμα πολιτικού διαλόγου που θα είναι ανοιχτός και επικοδομητικός μεταξύ των αραβικών κρατών του κόλπου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο σημείο, περιφερειακή διπλωματία. Στην έκθεσή μας επιμένουμε στο σημαντικό ρόλο που παίζουν τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του ΚΟΛ που διαμεσολάβησε με τους Παλαιστινίου στο πλαίσιο της κρίσης ε, στο Λίβανο, καταπολέμηση τρομοκρατίας και το Συμβούλιο Συνεργασίας του ΚΟΛ που πρέπει να πούμε ότι είναι και ένα παράδειγμα σταθερότητα στην περιοχή και μπορούμε να υπογραμμίσουμε τη βούληση του Συμβουλίου για να επικρατήσει η ειρήνη σε αυτή την ιδιαίτερα σταθή περιοχή. Αυτό ήδη το είχαμε και στην πρώτη έκθεση και καταλήξαμε με τους γιώδεις εισηγητές σε εξαιρετικές συμβαστικές προτάσεις για να μπορέσουμε να τονίσουμε αυτά τα στοιχεία. Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου είναι ένας πρώτης γραμμής εταίρος στην περιοχή. Έχει υπογράψει μάλιστα πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, μέσω της ε, Ισλαμικής ε, Τράπεζας Ανάπτυξης ε, μια συμφωνία με την Ήμρα για να χρηματοδοτηθούν σε ύψος 6 εκατομμυρίων δολαρίων κάποια έργα που θα πρέπει να γίνουν στη Γάζα πάρα πολύ επίγοντα και αυτό ζητάμε και με τη συμβαστική πρόταση 8. Αλλά βέβαια θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα 6 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό δεν επαρκεί, δεν αντιστοιχεί στις ικανότητες, στις οικονομικές των κρατών μελών. Ο διαθρησκιακός διάλογος τώρα και η αλαμιβαία κατανόηση. Η περιοχή των κρατών του κόλπου, των αραβικών κρατών του κόλπου αυξάνεται συνεχώς. Σε πολλές τροπολογίες με θυμίζεται ότι αυτά τα κράτη μπορούν και οφείλουν να διαματίσουν έναν επικοδομητικό ρόλο στο διαθρησκιακό διάλογο και μεταξύ Σιητών και Σουνιτών και όχι μόνο μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Πρόκειται για δικαιώματα τα οποία υπογραμμίζουν οι τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν. Τώρα, ο διαπολιτισμικός διάλογος επίσης τίθεται, όπως και τα διακυβεύματα για μια μεγαλύτερη αλληλοκατανόηση. Προτείνονται δύο επιλογέ. Πρώτα απ' όλα ανταλλαγέ πανεπιστημιακέ, που θα πρέπει να είναι πιο πυκνέ με μεγαλύτερη κινητικότητα εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού φοιτητών, μαθητών. Προτείνουμε επίση καλύτερη συνεργασία στον τομέα τη πληροφόρηση και επίση ενίσχυση σχεδίων όπω το Αλζίσρ. Γέφυρα θα πει για τη διπλωματία και τις δράσεις ευαισθητοποίησης. Σε ό,τι αφορά τώρα την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ρόλου των, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να βαθύνουμε τις σχέσεις αυτές, μέσω των τροπολογιών και των συμβιβασμών κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, προτείνουμε κάποιες επιλογές. Ξέρουμε ότι πλέον έχει διπλωματική υπηρεσία η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία πρέπει να αξιοποιήσει θα θέλαμε νέες διπλωματικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να προσθεθούν στη μία μόνο που υπάρχει, μία μόνο αποστολή υπάρχει, μέτρα το Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ορατότητα, δεν προβάλλεται στις χώρες αυτές του κόλπου και προς το παρόν δεν ε, διαθέτει τους σπόρους προς τούτο. Αν όμως θέλουμε να συμφωνήσουμε και να υπογράψουμε την υποδιαπραγμάτευση αυτή για τόσα χρόνια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις χώρες του κόλπου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη προβολή, να είναι πιο ορατή. Διμερείς σχέσεις τέλος είναι ένα ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Είχα πολλές συναντήσεις με τους κοιόδης εισηγητές. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε αν οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μείνουν σε αδιέξοδο για ακόμη μερικά χρόνια και κάποιοι πιστεύουν και συμμερίζομαι την άποψή τους αλλά και όλες οι πολιτικές ομάδες δεν συμμερίζονται ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, πολυμερή συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Συνεργασίας ε, του Κόλπου αν λοιπόν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε ή να ενθαρρύνουμε την σύναψη δημερών σχέσεων μεταξύ δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση και καθενός μεμονωμένου κράτου μέλου του Συμβουλίου Συνεργασία του ΚΟΛΠ. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε στι συναντήσει μα στην Επιτροπή αλλά και στη Συνδρία Ολομέλεια. Εν τέλει, δεν φαίνεται καμία μεμονωμένη περίπτωση στην έκθεση αυτή, γιατί στόχος της έκθεσης είναι να αναλύσει τις σχέσεις μας με το σύνολο ένα σύνολο, γιατί περί αυτού πρόκειται το Συμβόλιο συνεργασία του Κόλπου είναι ένα σύνολο και δεν θέλουμε να στοχοποιήσουμε ή να αναφέρουμε συγκεκριμένα κάποιο μεμονωμένο κράτος μέλος. Βέβαια, κάθε φορά που αναφέρεται σε τροπολογία ε, ένα κράτος συγκεκριμένο, εγώ προσπαθώ η τροπολογία αυτή να ενταχθεί σε ένα συμβιβασμό ώστε να διαγραφεί η άμεση μνήα, η απευθείας μνήα σε ένα κράτος μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Τέλος, μια διευκρίνηση έχει γίνει ένα μεταφραστικό σφάλμα, πολύ σημαντικό, από τα γαλλικά προς τα αγγλικά. Στην παράγραφο 4 συγκεκριμένα. Droit travail λέγεται στα, στο γαλλικό κείμενο. Labor law και όχι right to work πρέπει να είναι η μετάφραση στα αγγλικά γιατί μιλάμε για το εργατικό δίκαιο και όχι για το δικαίωμα προς εργασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μποντισλιο Πρόεδρος. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Ρίτσαρντ Howitt. Um, Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Μποντής ενδιαφέρεται για την περιοχή αυτή πολύ και διαπραγματεύτηκε με τους σκιώδεις με τρόπο δίκαιο και ολοκληρωμένο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να ε, επιτύχουμε συμβιβασμούς. Εμείς ε, θέλαμε να τονίσουμε την παράγραφο 6 και την αιτιολογική σκέψη Β όσον αφορά την ασφάλεια, ε, θέλαμε επίσης ε, ε, να πούμε ότι θέλαμε το Ισλαμικός να μην ακολουθεί την τρομοκρατία σαν επίθετο. Είμαστε απολύτως κατά της τρομοκρατίας, αλλά δεν χρειάζεται να βάζουμε τέτοιου είδους ταμπέλες Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα γλώσσας ε, και κατανόησης ε, της ε, μειονότητας και των μειονοτήτων και θέλουμε λοιπόν να αναφέρεται η λέξη μειονότητα στην παράγραφο 4. Είχαμε μία πολύ καλή συζήτηση όσον αφορά την, τις εκτελέσεις, την θανατική καταδίκη και το πώς θα ορίζαμε τις ε, την ε, θανατική καταδίκη. Και επομένως τώρα έχουμε μια, έναν πλήρη κατάλογο ε, και χαιρόμαστε πάρα πολύ και νομίζω ότι καλύτερα καταδεικνύουμε την αντίθεσή μας στην θανατική ποινή εάν αναφερθούμε σε κάποιους από τους τρομακτικούς τρόπους με τους οποίους αυτή εκτελείται ειρηνευτικές διαδικασίες. Ναι, θέλουμε ε, να στηρίξουμε αυτά που λέει ο κύριος Μποντή. έτσι ώστε στα κατεχόμενα να μπορεί να βοηθήσει ε, η βοήθεια, να φτάσει η βοήθεια της, είπε Όσον αφορά τώρα την τροπολογία μας 68 ε, ακόμα εκρεμεί, αφορά την εκπαίδευση και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Και τέλος, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο περίπλοκο σημείο. Θέλω να πω και στον κύριο Μποντής και στους υπολείπους ότι στην ομάδα μου μας απασχολεί πάρα πολύ σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες του κόλπου πολυμερός. Και θα θέλαμε κάπου να αναφερθεί ίσως εν είδη προσθήκης την επιθυμία μας για πολυμερείς συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει πραγματικά να υπογραμμίσουμε, να επιμείνουμε σε αυτήν την πολυμερή διάσταση των συμφωνιών. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι για μας είναι πολύ σημαντικό θέμα. Γι' αυτό το λόγο συμφωνούμε με τον εισηγητή αλλά θέλουμε να αλλάξει ο συμβιβασμός για την τροπολογία 24. Ε, ε, η κυρία Κιμάκη έχει μία ε, τροπολογία η οποία θέλουμε να ψηφιστεί χωριστά. Δεν ξέρω αν είναι εδώ η κυρία Κιμάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να ζητήσω και από τις άλλες ομάδες να μας ακολουθήσουν. Πάντως, να υπογραμμίσω ότι η συζήτηση ήταν πάντα πολύ συνενετική και ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Ευχαριστούμε. Η κυρία Πρίμπολς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, των Πρασέινων θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μποντή, τον εισηγητή για το γεγονός ότι ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστη και ανοιχτή η συνεργασία με τους κοιόντες εισηγητές. Έχουμε πλέον κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες προετοίμασε και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα νομίζω ότι το κείμενο θα καταλήξει να είναι πολύ ισόρροπο. Από πλευράς όμως της ομάδας μου θεωρούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των ε, ε, οργανώσεων πολιτών και την επικύρωση διεθνών συμβάσεων από τις εμπλεκόμενες χώρες. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και οι έξι χώρες του κόλπου έχουν ε, μοναρχία και μάλιστα κληρονομική με περιορισμένη συμμετοχή ιδιαίτερα των γυναικών και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν καν εκλεγμένα κοινοβούλια. Θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση λείπει, υπάρχει έλλειψη διεθνούς ε, προστασίας και ελέγχου σε ό,τι αφορά τις ε, διεθνείς συμβάσεις και τον διεθνή έλεγχο. Έχω κυρίως υπόψη μου τη συνθήκη σε ό,τι αφορά την κατάργηση διακρίσεων κατά των γυναικών, την διεθνή συνθήκη σε ό,τι αφορά τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα, διεθνή συνθήκη για την οικονομική, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα και τέλος ε, ε, η συνεργασία με τις θεματικούς μηχανισμούς, του τομεακούς μηχανισμούς του ΟΗΕ οι οποίοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα επίσκεψης και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ε, δικηγόρων και των νομικών. Η έκθεση θα πρέπει να παρατρύνει τις χώρες του κόλπου, να εγκρίνουν τις συμβάσεις αυτές και να επιδιώξουν μεγαλύτερη συνεργασία με τις ε, αρχές του ΟΗΕ, το οποίο ασφαλώς θα ωφελήσει και τον λαό της κάθε χώρας και προς αυτή την κατεύθυνση έχει υποβάλει η ομάδα μου κάποιες τροπολογίες, τις οποίες και ελπίζω να υποστηρίξετε. Τέλος, Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, διαπιστώνω ότι η Επιτροπή Ήτρε σε μία από τις τροπολογίες της προτείνει η συνεργασία με τις χώρες του κόλπου σε τομέα, ε, στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας να ενισχυθεί. Προτείνω να ακολουθήσουμε την γνωμοδότηση αυτή και το ίδιο επιδιώκει και η τροπολογία 62 της ομάδας μου. Ελπίζω να εγκριθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάιερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η δική μου πολιτική ομάδα θέλει επίσης να ευχαριστήσει τον κύριο Ποτίσα ε, για τη δουλειά που έχει κάνει. Εμείς ωστόσο Λόγω των γεγονότων ε, της Τίνιδας αλλά και της Αιγύπτου ε, σκεπτόμαστε σε ποιο βαθμό, ε, μέχρι ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δρομολογήσει όλους τους μηχανισμούς και να κινητοποιήσει όλο το δυναμικό είτε για να συνοδεύσει είτε για να καταγγείλει, να παρακολουθήσει μάλλον είτε για να καταγγείλει όλες αυτές τις, την κακομεταχείριση θα έλεγα κατά του πληθυσμού και των γυναικών. Είδαμε τι έγινε σήμερα στην πλατεία ανεξαρτησίας του Καΐρου. Πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα ήταν εκεί. Αν έπρεπε να αξιολογήσουμε και να πούμε σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια επιρροή εμείς ως ομάδα πολιτική νομίζω ότι πολύ λίγο επηρεάζουμε και πολύ λίγο χρησιμοποιούμε και τους μηχανισμούς καλής γειτονίας. Δεν τους χρησιμοποιούμε για να παρακολουθήσουμε και για να ενισχύσουμε, να τονώσουμε τον εκδημοκρατισμό ε, είτε φεουδαρχικών ε, μονοπωλίων είτε τυραννιών ε, που έχουν εγκαθιδρυθεί στην περιοχή αυτή του κόσμου. Έχουμε λοιπόν αυτήν την έννοια υποστηρίξει και υποβάλει σημαντικές τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα για να πούμε ότι εμείς είμαστε ιδιαίτερα ιδιαίτερα ε, επιφυλακτική και αρνητική στο να υποκατασταθεί η ουσία ε, της όλης αυτής της υπόθεσης με μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που δεν θα λαμβάνει υπόψη ε, τις ασυμμετρίες. Δεν είναι τα πάντα εμπόριο, ούτε πρέπει να είναι όλα ελευθερία αγοράς, μια ασαρρύθμιση της άναρχης αγοράς, έχοντας υπόψη και τη χρηματοπιστωτική κρίση που βιώνει και η Ευρώπη και ο υπόλοιπο κόσμος. Υποβάλαμε λοιπόν διάφορες τροπολογίες, πρώτα απ' όλα για να προσπαθήσουμε να δούμε ένα συγκεκριμένο προφίλ για αυτή την τόσο σημαντική γεωγραφική περιοχή. Ξέρετε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε από τότε που αποφάσισε ε, η ενεργειακή της εξάρτηση να αποτελέσει εθνικό πρόβλημα και μετά από αυτή τη διακήρυξη συγκεκριμένη περιοχή είναι είναι ε, μία ζώνη μόνιμου επανεξοπλισμού και δεν νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το ενστερνιστεί και να το ασπαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το αντίθετο και πρέπει να ζητήσει αφοπλισμό μια περιοχή η οποία πρέπει και μπορεί να διδραματίσει ένα σημαντικό ε, ε, ρόλο και απέναντι προ το Ιράκ και προ το Ιράν και προ την Εγγύη Ανατολή. Έχουμε και μία πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΙΠΑ και Σαουδική Αραβίας, στρατιωτικέ βάσει στο Μπαχρέιν, στο Ομάρ, στην Σαουδική Αραβία. Άρα ο ρόλο που παίζουν αυτέ οι βάσει των ΙΠΑ σε σχέση με συγκρούσεις όπως αυτή του Ιράκ μας οδηγούν στο να υποβάλουμε τροπολίες ακριβώς ε, ώστε από τη δική μας την πλευρά ως Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση τα χαρακτηριστικά μας να πρέπει να κυριαρχούν οι προθέσεις μας για ε, προοδευτική αποστατικοποίηση της περιοχής και ενεργειακή εξάρτηση δεύτερον στην προκειμένη περίπτωση βέβαια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τον είπα να μην μετατραπεί σε ένα πρόβλημα ασφαλείας. Οι ενεργειακές εξαρτήσεις πρέπει να επιλύονται με δια της διπλωματικής οδού. Ποτέ δεν θα πρέπει να αναπτύσσονται στρατιωτικές δυνάμεις δυνάμεις εκτός των ε, εδαφών μας, εκτός επικρατείας μας. Και βέβαια εδώ λέμε ότι κατά καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας όπως πράττουμε οι πολιτισμένες, όπως θα έπρεπε να πράττουμε οι πολιτισμένες χώρες. Όχι βομβαρδίζοντας από 10.000 μέτρα αθώους ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν υποβάλει τις τροπολογίες μας Πιστεύουμε ότι στόχος τους είναι να κάνουν αυτή την ανεξάρτητη αναφορά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στάση που πρέπει να έχει απέναντι στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν τροπολογίε επίση, τι οποίε ε, θα τι υπερψηφίσουμε γιατί είναι κατά τη διάκριση μεταξύ των δύο φύλων, καταγγέλουν την κατάσταση των γυναικών στι χώρε αυτέ, είναι υπέρ τη ε, πρόθεση, τη ελευθερία, τη έκφραση, τη ανεξιθρησκεία, τη κατάργηση τη θανατική ποινή. Ζητούν επίση καλύτερη μεταχείριση των εργαζομένων που είναι μετανάστε και προέρχονται από τρίτε χώρε και επίσης ε, μείωση του εμπορίου όπλων και εξοπλισμών. Θα δούμε πώς θα προκύψει το, το τελικό κείμενο, ποια μορφή θα έχει και θα δούμε ανάλογα πώς θα, θα κινηθούμε, αν θα το στηρίξουμε ή όχι. Κυρία Γιατεμάκη, το λόγο. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, του κύριο Μποντή, για την εξαιρετική έκθεση και για την εξαιρετική συνεργασία. το κείμενο εντοπίζει τους προβληματικούς τομείς αλλά και τις ευκαιρίες που ενέχει η σχέση μεταξύ Ευρώπης και των χωρών του κόλπου. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ε, συνεργασίας του κόλπου. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Βόρεια Αφρική, για παράδειγμα, καταδεικνύουν ότι η Ευρώπη και οι χώρες αυτές έχουν όντως τομεί κοινή ε, κοινών συμφερόντων και σε τομεί εξωτερική πολιτική. Αναπτύσσοντα λοιπόν τι σχέσει αυτέ, συμβάλλουμε στην ε, περιφερειακή συνεργασία που είναι απαραίτητη για τις σχέσεις καλής γειτονίας και σταθερότητας στην περιοχή. Επιπλέον, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρήκαμε πόσο σημαντική είναι η παιδεία και οι ανταλλαγέ φοιτητών. Και το τονίσαμε αυτό. Η βάση για την μελλοντική συνεργασία θα πρέπει να βασίζεται στην νεολαία της Ευρώπης. Και θα ήθελα τέλος να απαντήσω στον συνάδελφο Χαουίτ, ο οποίος ρώτησε περί διμερής συνεργασίας. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να βελτιωθούν οι διμερείς σχέσεις με τις χώρες του κόλπου. Τονίζω και υπογραμμίζω επίσης πόσο σημαντικό είναι να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς την ύπατη εκπρόσωπο, αντιπρόσωπο, την Κάθριν Άστον, για την εντατικοποίηση των σχέσεων με τις χώρες του κόλπου. Οι χώρες είναι διαφορετικές, έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και είναι καλό να λαμβάνουμε πληροφορίες από κάθε χώρα για τις ανάγκες της και τις προτεραιότητές τους. Ευχαριστώ κύριε Σλαφράγκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρει κανείς έναν καταλληλότερο για την έκθεση αυτή συγκεκριτή από τον κύριο Ποντή. Θέλω να χαιρετήσω τον συγκεκριτή για την εξαιρετική του δουλειά, για την υποβολή τη έκθεση αυτή, που πραγματικά περιλαμβάνει όλα τα σοβαρά ε, σημεία τα οποία μα ενδιαφέρουν ε, στο πλαίσιο τη σχέση μα με τι χώρε του Συμβουλίου Συνεργασία του Κόλπου. Πιστεύω ότι πράγματι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ε, δημιουργία μια στρατηγική σχέση με τι χώρε αυτέ που θα ενσωματώνει πολλά από τα στρατηγικά ζητήματα τα οποία αναφέρονται και στην έκθεση. Αυτό το οποίο θέλω εγώ να πω έξω, άμα το συζητήσουν πολιτική ομάδα, είναι ότι εμεί πράγματι πιστεύουμε ότι υπάρχουν ευεργετικέ επιπτώσει μέσα από μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος που θεωρεί ότι το εμπόριο είναι πρόοδος, είναι ειρήνη. Όταν κάποιες από τις ανταγωνιστικές χώρες έχουν πιστεί ε, ότι αυτό ισχύει, ε, εμείς ε, δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα σύνορά μας. Σήμερα με τις χώρες Μερκοσού συζητήσαμε για την συμφωνία αυτή που θα πρέπει να επιδιώκει ισορροπία μεταξύ της, του ανήκει σε μια ομάδα όπως παραδείγματος χάρη η ΚΑΠ και η συνεκτικότητα και συνέπεια με τους στόχους μας. Θέλουμε να έχουμε μία ισορροπία. Πρέπει να εφαρμόζουμε τις αρχές μας με συνέπεια και ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε και τα συμφέροντα αυτού του κλαμπ, Αυτή της ε, σχέσης. Εκεί πρέπει να βρούμε την χρυσή τομή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό και η υπηρεσία εξωτερική δράση να αναπτύξει τι δραστηριότητέ τη για να είναι μεγαλύτερη όλο και περισσότερο προβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή του κόλπου. Και επίση η κίνδυνη που μπορεί να εγκυμονεί ε, μια κλιμάκωση, ε, αύξηση των εξοπλισμών, είναι κάτι το οποίο αναφέρει και ο εισηγητής μα στην παράγραφο 6. Τώρα, σε ό,τι αφορά την θεμητή, την νόμη ανησυχία για την κατάσταση της Βορείου Αφρικής, βλέπουμε να επεκτείνεται γενικότερα στον αραβικό κόσμο και αυτό πρέπει να αναφερθεί στην έκθεση. Το λέει πολύ σωστά ο εισηγητής στο σημείο 4 νομίζω, όπου καλεί τις χώρες ε, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου ε, να προχωρήσουν πέραν από, ε, μάλλον να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και να προωθήσουν περισσότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα. και έτσι πιστεύουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση και μάλιστα σημαντικά. Δεν έχω πολλές παρατηρήσεις να κάνω. Νομίζω ότι η αναφορά στην ενεργειακή συνεργασία είναι μια θεμελιώδης αναφορά λαμβάνοντα υπόψη την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και το πόσο επηρεάζει αυτό την οικονομική κατάσταση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, πολύ αποφασιστική σημασία έχει η εκπαίδευση και νομίζω ότι η έκθεση πηγαίνει προς την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μόνη σύσταση που έχω να κάνω προς ε, τον εισηγητή συμφωνώ βέβαια με όλα όσα αναφέρει, είναι όταν μιλάει για αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση, για αυτή τη στρατηγική σύνδεση, να αναφερθεί στα ανθρώπινα δικαιώματα λέγοντας ότι θα πρέπει να βασίζεται στις αξίες και στις αρχές που εμπνέουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είδαμε η ανάπτυξη μιας realpolitik ε, στη βόρεια όχθη της Μεσογείου, το μόνο που έφερε δεν ήταν ούτε, μάλλον δεν έφερε ούτε περισσότερη σταθερότητα, ούτε περισσότερη ευημερία, ούτε περισσότερη δημοκρατία και όπως μιλάγαμε παρουσία και του Επιτρόπου Φίλε, νομίζω ότι πρέπει να αντιλήσουμε κάποια διδάγματα, όχι να αναζητήσουμε ενόχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν πρόκειται περί αυτού, απλά οι διχόνοι του παρελθόντος να προσπαθήσουμε να γίνουν ε, η ομόνια και η αρμονία του παρόντος και του μέλλοντος. Άρα όχι μόνο αναφορά στο σημείο 4 στα δικαιώματα αλλά και στις αξίες της Ένωσης. Παναλαμβάνω ότι ο εισηγητής μας είναι ειλικρινά ένας εισαγητής ε, που δεν θα μπορούσε να βρει ε, αντάξιο ε, στις γνώσεις και στην εμπειρία για να πραγματευτεί αυτό το θέμα. Κύριε Μποντής, θέλετε να πείτε κάτι, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι άκουσα με ιδιαίτερη ευαισθησία τις παρεμβάσεις εκτιμώ και εγώ ε, τις προσπάθειες ε, και τη συνεργασία των σκιωδών εισηγητών για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Θα είμαι σύντομος λοιπόν στην παρέμβασή μου. Μετά και από τα λόγια του κυρίου Σάλα ε, που πολύ ε, επιμείναμε σε αυτό το κείμενο και πολλές τροπολογίες είχαν ως στόχο ακριβώς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κεντρικό στοιχείο των σχέσεών μας ε, με αυτή την περιοχή του κόσμου. Ωστόσο, μετά από την παρέμβαση του κυρίου Μάγερ, ε, θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν είναι η ίδια σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες ε, της Μεσογείου έχουν αδιαφορετικέ σχέσεις μεταξύ του στο πλαίσιο συμφωνίας γειτονία. Όταν έχουμε να κάνουμε με τι αραβικέ χώρε του κόλπου, δεν είμαστε στα ίδια πράγματα. Δεν έχουμε καν συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Αυτό ε, που λέω τώρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε κατά μέρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά είναι προφανέ ότι το επίπεδο απαιτήσεων που μπορεί να έχουμε δεν μπορεί να είναι το ίδιο με ένα σύνολο κρατών με τα οποία εδώ και 20 χρόνια διαπραγματευόμεθα μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και να είναι ίδια, επαναλαμβάνω, με χώρε όπω η Αίγυπτο ή Τινησία, χώρε με τι οποίε έχουμε συμφωνίε σύνδεση, στι οποίε ρητό αναφέρεται η ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρία Μπρίπολ, πολύ σωστά είπατε ότι αυτά τα κράτη είναι ένα από τα κοινά του χαρακτηριστικά, όλα τους, είναι κληρονομικέ μοναρχίε. Πράγματι, όταν του κάναμε τη σχετική παρατήρηση, μα είπαν «Μα και εσεί έχετε πολλέ μοναρχίε στην Ευρώπη, κληρονομικέ μοναρχίε. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι η ίδια οργάνωση εξουσία, αλλά πρέπει να παρατηρήσουμε ότι και στην Ευρώπη υπάρχουν μοναρχίε. Τώρα, θανατική ποινή. Γίνεται πολλή λόγο. Δεν μιλάμε για τη μοναρχία, μιλάμε για τη θανατική ποινή και μιλάμε και για ε, τους ακροτηριασμούς ο κολλασμού αξιόπινων πράξεων. Και επιμένουμε, μένουμε σε αυτό συνεχώ. Τώρα, αφοπλισμό. Ο κύριο Μάγκερ έθεσε το θέμα αυτό. Πράγματι, θα είμαστε όλοι μας πολύ πιο ήσυχοι, πολύ πιο ήρεμοι και γαλήνοι αν είχαμε έναν αραβοπερσικό κόλπο που θα ήταν αποστρατιωτικοποιημένο. Αλλά όταν μιλάμε για αποστρατιωτικοποίηση τη αραβική όχθη, δηλαδή Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, εγώ σκέφτομαι λίγο τα λόγια το Φρανσουά Μιτερά στην Bundestag που έλεγε στην Ευρώπη οι πύραυλοι είναι στη, στην Ανατολή και οι, φιλιρινιστές είναι στην ε, Δύση. Ε, κοιτάξτε, δεν μπορούμε προκλητικά να ζητούμε ε, αφοπλισμό της αραβικής όχθης σε μια περιοχή που δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα, αυτή την άσκηση αφοπλισμού. Τώρα, αν δούμε εκ παραλίλου τι γίνεται στο Μαγκρέμπ και το συγκρίνουμε με αυτά που γίνονται στον κόλπο, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια όρια σε αυτή την άσκηση. Είναι λίγο αντιφατικές αυτές οι καταστάσεις. Για παράδειγμα, σε ένα από τα κράτη-μέλη, το Κατάρ, του Συμβουλίου Συνεργασίας ε, του Κόλπου, έχουμε το Αλτζαζίρα, το σταθμό αυτό, που από γενικής, ε, κατά τη γενική ομολογία ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία του επαναστατικού κινήματος ε, και της επανάστασης εξέγερσης χθες στην Τινησία σήμερα στην Αίγυπτο και έχετε στο ίδιο κράτος ακριβώς, το Κατάρ, 500 μέτρα από το Αλτζαζίρα έχετε το κέντρο διοίκησης των επιχειρησιακών, αμερικανικών επιχειρησιακών δυνάμεων στον κόλπο. Επομένως, υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Θα μπορούσε να πει κανείς και για σχιζοφρένεια στην εξωτερική πολιτική κάποιων κρατών που από τη μία ενθαρρύνουν επαναστατικά κινήματα αλλά αποτελούν βάση ε, της παρουσίας των Αμερικανών στον κόλπο από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, δεν μπορούμε έτσι πολύ εύκολα να αφήσουμε κατά μέρο το θέμα τη θανατική ποινή, των ακροτηριασμών, τη διαφορά ε, μεταξύ των δύο φύλων, της ανισότητα, της κατάστασης των οικονομικών μεταναστών, ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν θέλουμε να δώσουμε απ' την άλλη όμω και την εντύπωση ότι θέλουμε να επιβάλλουμε ένα πολιτικό μοντέλο γιατί και είπα και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θέλησαν το 2003 να επιβάλλουν ένα πολιτικό μοντέλο στον κόλπο. Είχαμε το δεύτερο πόλεμο του Ιράκ. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε. Άρα πρέπει και να είμαστε κατηγορηματικοί απέναντι στις αρχές μας, αλλά να είμαστε και λίγο μετριοπαθείς και μετριόφρονες σε σχέση με κάποιες πολιτικές ε, που εφαρμόζει η Δύση σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να πω ότι θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 10 Φεβρουαρίου για την έκθεση αυτή. Και περνάμε λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα στην έκθεση του κυρίου Μπροβέρα, του Αντιπροέδρου, για τα μεταναστευτικά ρεύματα που προκύπτουν από την αστάθεια. Στόχος και ρόλο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα θέμα το οποίο είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο παραποτέ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δόκιμη η στιγμή στην οποία έρχεται η έκθεση αυτή και να ευχαριστήσω αμέσως τους συναδέλφους ε, που προτίθενται να ασκήσουν είτε κριτική είτε να προσθέσουν κάποια σημεία. Η μετανάστευση είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα πολύ συχνά, υπερβολικά συχνά ε, στηρίζεται σε προκαταλήψεις και ρυθμίζεται από υποκειμενικές ε, θεωρήσεις που εμποδίζουν την αντικειμενική θεώρηση, πράγμα που εμποδίζει βεβαίως με τη σειρά του τον καθορισμό σωστών πολιτικών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο λοιπόν το οποίο ε, πήρε πολύ σημαντικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια με αντίκτυπο όχι μονάχα οικονομικό ε, ή ε, πολιτικό αλλά ανθρωπιστικό, κοινωνικό κλπ. Υπάρχει η νόμιμη μετανάστευση, υπάρχει και η παράνομη μετανάστευση ο λόγος ε, για τον οποίο κάποιος ε, μεταναστεύει ε, είναι είτε πολιτικές καταστάσεις, είτε φυσικές καταστροφές, είτε καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έλλειψη δημοκρατίας, αλλά κατά κύριο λόγο μεταναστεύουν οι άνθρωποι γιατί επιθυμούν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και θέλουν να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η λαθρομετανάστευση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ε, το γεγονός δηλαδή ότι είναι λαθρέοι οι άνθρωποι αυτοί ε, οδηγεί σε μία, ε, στην μαύρη εργασία, οδηγεί σε μία κατάσταση νέας σκλαβιάς που πιστεύαμε ότι έχει πλέον ε, περάσει στη σφαίρα του παρελθόντος αλλά δυστυχώς ε, βλέπουμε ότι ε, ξαναρχίζει και βεβαίως έχουμε σαν παρεμπίπτον φαινόμενο τις κακουχίες, την βία, τη σεξουαλική βία ακόμα και την τρομοκρατία. Πιστεύω ότι η παράνομη μετανάστευση δεν αντιμετωπίζεται μονάχα με σαφείς, έστω και αν αυστηρούς νόμους, ε, ούτε μόνο με την καταστολή ή την απομάκρυνση, αλλά χρειάζεται, είναι απαραίτητο να έχουμε μια αποτελεσματική και γενναιόδορη συνεργασία με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι, οι άνθρωποι αυτοί, οι μετανάστες. Πολιτικές λοιπόν συνεργασίας, όχι σαν αυτές του παρελθόντος που απέτυχαν. 50 χρόνια μετά βλέπουμε τα αποτελέσματα ενώπιόν μας. Βλέπουμε ότι δεν βοηθούμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και το μεταναστευτικό ρεύμα αντί να μειώνεται αυξάνεται και πρέπει να κατανοήσουμε τα αίτια της αποτυχίας ε, εάν θέλουμε να ε, προχωρήσουμε επιτυχώς προς το μέλλον. Η αποτυχία οφείλεται στην ε, διαφθορά και στις διαρθρωτικές δυσκολίες που παρουσιάζουν οι χώρες προέλευσης. Επίσης, από το ότι οι χώρες δωρητές ασχολούνται με θέματα τα οποία δεν είναι απαραίτητα πρώτης ανάγκης ε, για τις χώρες προέλευσης μια συνεργασία, μια καθαρά αναπτυξιακή συνεργασία, όμως έστω και αν ήταν τέλεια δεν θα μπορούσε να απαντήσει σε ένα τόσο περίπλοκο ε, και με τόσες πολλές αποχρώσεις φαινόμενο. Το κυρίαρχο πρόβλημα είναι η αστάθεια η αστάθεια η οποία μπορεί να είναι πολιτική, μπορεί να είναι οικονομική, μπορεί να οφείλεται σε φυσικά αίτια, σε φυσικές καταστροφές, αλλά ε, και σε πολιτικούς λόγους. Ε, και αυτό το καταλαβαίνουμε πολύ καλά βλέποντας τι συμβαίνει στην Τινησία, στην Αίγυπτο, στη Βόρεια Αφρική, στις χώρες Μαγρέμπ. Θα μπορούσα να πω ότι σε γενικές γραμμές η πολιτική αστάθεια αφορά ε, συνήθως ε, μεγάλες ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πολύ συχνά οφείλονται σε αβάναυσες δικτατορίες. Η οικονομική αστάθεια οφείλεται στις μεγάλες διαφορές αποκλήσεις ανάμεσα στον Παρά και τον Νότο. Η δε κατηγορία των περιβαλλοντικών ας πούμε, φυσικών προβλημάτων είναι αυτά τα μεγάλα φυσικά φαινόμενα, τα ακραία φυσικά φαινόμενα, οι φυσικές καταστροφές που οδηγούν σε εκτοπισμό μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Ας μιλήσουμε καλύτερα για την σταθερότητα και όχι την αστάθεια. Πιστεύαμε πάντα ότι η πολιετής διακυβέρνηση Μουμπάρακ στην Αίγυπτο θα οδηγούσε σε κάποια ε, σταθερότητα που θα ήταν πολιτική και η οποία όμως κατέρευσε σαν τραπουλόχαρτο γιατί μέσα στα πλαίσια αυτής ε, της εξέγερσης στο Μαγκρέμπ ε, βλέπουμε ε, σαν βάση την κοινωνική αστάθεια και επομένως αυτή η ηρεμία που βλέπουμε στον πολιτικό κόσμο ήταν ηρεμία επιφανειακή και στην Τινησία όπου η κατάσταση ήταν διαφορετική από ό,τι στην Αίγυπτο αλλά και στην Αίγυπτο και στην Αλγερία κλπ αυτό που λείπει τελικά είναι αυτή η δομή ε, κοινωνικής ε, ε, διαβούλευσης, διαβούλευσης μεταξύ των πολιτών έτσι ώστε τα αιτήματά τους να αναφέρονται στην κυβέρνηση. Αναφέρομαι εδώ στο, στο συνδικαλιστικό κίνημα, αναφέρομαι επίσης στα πραγματικά πολιτικά κόμματα, στα πλαίσια των οποίων μπορεί κανείς όντως να διαεξάγει πολιτική συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών. Αναφέρομαι επίσης στην δυνατότητα του συνεταιρίζεστε, στην δυνατότητα της δημιουργίας οργανώσεων και ενώσεων, όλων αυτών δηλαδή των δομών που επιτρέπουν στον λαό να ζουν εν δημοκρατία και να εκπροσωπούν δημοκρατικά τα δικαιώματά τους. Επομένως αυτή ε, η τύπη σταθερότητα ε, πολιτική σταθερότητα, κυβερνητική σταθερότητα δυναμητίζεται από την έλλειψη κοινωνικών υποδομών ε, και διαρθρωτικά οργανωμένων θεσμικών οργάνων και οργανώσεων που θα δημιουργήσουν πραγματικά ε, την βάση για ε, πραγματική πολιτική σταθερότητα. Η οικονομική, η δημοσιονομική βοήθεια βεβαίως είναι απαραίτητη όμως θα πρέπει να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να απαντά σε συγκεκριμένα αιτήματα ε, των πληθυσμών στους οποίους ε, ε, αναφέρεται μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ε, υποστήριξης αλλά και παρακολούθησης των χωρών που προτιθέμεθα να στηρίξουμε στήριξη έτσι ώστε να δημιουργήσουν αυτές τις κοινωνικές, πολιτικές και λοιπές υποδομές που οποιαδήποτε δημοκρατία χρειάζεται για να σταθεί στα πόδια της. Εγώ ε, κυρίως ε, μου είναι ιδιαίτερος προσφυλαίης η ιδέα των ίσων ευκαιριών, των ίσων δυνατοτήτων, μεταξύ άλλων βεβαίως, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μου είναι ιδιαίτερος προσφυλές. Αυτή ε, η ισοδικία, αυτή η δυνατότητα ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ όλων των πολιτών, θεωρώ ότι είναι βάση της δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να καλέσω τον κύριο Μπροκ, ο οποίος θέλει να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό, το θέμα της μετανάστευσης. And, uh, Mr. Uh, Και ο κύριος Τάνοκ μετά. Δεν ζήτησε το λόγο, Πρόεδρε. No, okay. Εντάξει τότε. Ο κύριος Τάλπτο για δύο λεπτά σκιώδης συζητητής. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι πρόκειται για ισορροπημένη έκθεση. Ο κύριος Προβέρα, ο εισηγητής, μας εξήγησε με μεγάλη λεπτομέρεια το τμήμα εκείνο Τη έκθεση που πραγματεύεται τι ροέ, τι μεταναστευτικέ που προέρχονται από ε, αστάθεια. Υπάρχει και άλλη μια διάσταση, ο ρόλος της ε, ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Οι ροέ. θα πρέπει να προσπαθήσουμε, στόχος μας να είναι να υπάρχει συντονισμένη δράση και να δίνεται βοήθεια υπό όρους. Φυσικά γίνεται εξαίρεση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Θα πρέπει να πω όμως ότι ο κύριος Προβέρα είχε ένα πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσει. Γιατί πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό μπλεκόμαστε και επικρατεί μια σύγχυση. Και γιατί? Γιατί μιλάμε για μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική για τη μετανάστευση. Ενώ δεν υπάρχει πολιτική, εγχώρια πολιτική, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να αποτυπώνει την πολιτική, τη μεταναστευτική στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει καν κοινή θέση από αυτού. Άρα ήταν δύσκολο το να βρεθεί ισορροπία για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Thank you. I'll be brief. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ, κύριε Προβέρα, για την εισαγωγή που μας κάνατε. Αναφέρθηκαν πολλά στοιχεία υπό ευρεία έννοια και πολλά ακόμα θα έχουμε να διευκρινίσουμε. Ελπίζω ως εισηγητές και όντες να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Θα ήθελα συγκεκριμένα να σας ε, ρωτήσω κατά πόσο θα αναλογιζόσαστε την εφαρμογή ενός συστήματος μπλε κάρτα για ε, ερευνητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αναφέρεστε σε μετανάστες σε άλλες χώρες, αναφέρεστε στην κατάσταση στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μεγάλο φάσμα μεταναστών και κάποιοι είναι μετανάστες γνώσης, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι πρέπει και αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους γιατί προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί πέρα από τα οικονομικά συμφέροντα προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους. Να σας ρωτήσω επίσης, επίσης αν σκοπεύετε να τονίσετε την πρόληψη της δημιουργίας μεταναστευτικών ροών, γιατί σε πολλά μέρη του κόσμου είναι σε πολύ ευάλωτη θέση οι μετανάστες. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα παιδιά. Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα θέματα τα οποία με ενδιαφέρει να μάθω την άποψή σα. Θα περιοριστώ σε αυτά επί του παρόντος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σέβεριν λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρε νομίζω ότι η έκθεση αυτή όχι μόνο είναι ισορροπημένη αλλά και σύνθετη, περίπλοκη. Ο εισηγητή προσπάθησε να περιγράψει τα φαινόμενα σε όλη του την πολυπλοκότητα. Τα φαινόμενα τη μετανάστευση. Να ήθελα να πω ότι μου άρεσε το ότι τονίστηκε ότι δεν είναι λύση και απάντηση η καταστολή. Δύο συγκεκριμένα στοιχεία. Καταρχάς, να επαναλάβω αυτά που ήδη είπε ο συνάδελφος Μοντάλγκο. Θεωρώ ότι θα πρέπει στην έκθεσή σας να επισέλθει ένα στοιχείο για να ενισχυθεί η ανάγκη σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής Μεταναστευτική πολιτικής της Ένωση και της εξωτερική πολιτικής της Ένωση για τη μετανάστευση. Τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω, αυτό που αναφέρεται ως brain drain, διαφυγή εγκεφάλων. Δεν μιλάμε μόνο για οικονομική αστάθεια, αλλά υπάρχει και η ανάγκη ανάπτυξης του κάθε ατόμου, το οποίο φυσικά μπορεί να είναι πολύ υποφελές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι πολύ επιζήμιο για τις χώρες προέλευσης. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί αστάθεια, το οποίο θα ενισχύσει τις μεταναστευτικέ ροές με νόμιμο ή παράνομο τρόπο. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να αφιερώσετε κάποια προσοχή και στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριο Στάνοκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια γενναία απόπειρα του κυρίου Προβέρα σε έναν ουδέτερο τόνο να απευθυνθεί και να πραγματευτεί ένα από τα πιο έντονα πολιτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στις ε, χώρες μας. Στην περιφέρειά μου του Λονδίνου η μαζική μη ελεγχόμενη μετανάστευση ύψους ίσως και 2 εκατομμυρίων, ε, εκατομμυρίων ανθρώπων αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες για τον κόσμο, για τους πολίτες μου. Α, συγγνώμη. Αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες, λοιπόν. Και ασκεί μία τεράστια πίεση, για παράδειγμα, στη Βρετανία, σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει που τίθονται και τις αξιώσεις που τίθονται για τις δημόσιες υπηρεσίες, για τα σχολεία και το καθεξής, σε ό,τι αφορά και θέματα ενσωμάτωσης. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο προφανώς πρέπει να το συζητήσουμε με ανοιχτό τρόπο, χωρίς όμως να προκαλούμε. Δεν αποδεχόμαστε στην ομάδα μου ότι η μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να καταστεί ε, ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και ένα από τους τομείς όπου θεωρώ ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να υπάρξει ευρωπαϊκή ενίσχυση προς φτωχε χώρε όπου υπάρχει μεγάλη ενεργία για παράδειγμα στου νέου, στο Μαγκρέμπ Νομίζω ότι έχουμε καθήκον να βοηθήσουμε στη σταθεροποίηση των χωρών αυτών και από πολιτική και από οικονομική άποψη και εν μέρη για να αποτρέψουμε την εκροή ε, μεταναστών προς τις χώρες μας. Και ίσως να χρηθεί απαραίτητη και η ανθρωπιστική βοήθεια. Νομίζω ότι στην Αφγανιστάν, στη Ζιμπάμπουε, οι Κούρδοι, όλες αυτές οι χώρες ε, έχουν στείλει πολλούς μετανάστες στις χώρες μας γιατί υπάρχουν άσχημες συνθήκες. Αν θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση θα πρέπει να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό που δεν μ' αρέσει είναι να συμπεριλάβουμε μια πολιτική επιλογή των καλύτερων όπως και το σύστημα της μπλε κάρτας για τους ε, επιστήμονες. Αυτό νομίζω ότι υπονομεύει και υποσκάπτει τις φτωχές αυτές χώρες και καταδικάζει τη χώρα σε ισόβια φτώχεια. Και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Και έτσι μοιραία δημιουργείται ένας ε, οικονομικός τέτοιος φαύλος κύκλος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αγκουράκης για δύο λεπτά. Μικρόφωνο. Ε, Τώρα θα τα πω στα ελληνικά. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, εμείς ε, διαφωνούμε κάθετα με την έκθεση ε, γιατί δεν θίγει το ουσιαστικό ζήτημα, την ουσιαστική αιτία και πολλές ουσιαστικές αιτίες που ε, έχουν ε, ως αιτία του το πρόβλημα της μετανάστευσης. Καταρχήν, νομίζω ότι όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά ο καπιταλιστικός κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση οικονομικής κρίσης και όπου το ζητούμενο είναι η συμπίεση του κόστου εργασίας, όπως ξέρετε, που είναι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόβλημα αυτό θα εντείνεται όλο και περισσότερο για τον πολύ απλό λόγο ότι οι μεγάλες πολυεθνικές στο μεγάλο κεφάλαιο θα θέλει πάντα φτηνή εργατική δύναμη και το μεταναστευτικό ρεύμα θα χρησιμοποιείται σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα, εάν δεν αναπτυχθεί μια άλλη πολιτική, αν δεν υπάρχει μια άλλη ανάπτυξη με γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων και όχι το καπιταλιστικό κέρδος, πάντα θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα και θα εντείνεται με κάθε μέρα που περνάει. Δεύτερο ζήτημα, πολύ σημαντικό, είναι ότι δεν αναφέρονται οι τεράστιες ευθύνες του δυτικού κόσμου, του κόσμου της εκμετάλλευσης και των πολυεθνικών που ε, ανταγωνίζονται για αγορές, που ανταγωνίζονται για σφαίρα επιρροής, που ε, προκαλούν ε, πολέμους και αστάθεια και αυτό είναι ένα από τα βασικότερα ε, μεταναστευτικά ρεύματα που υπάρχουν σήμερα. Δεν είναι δυνατόν κύριε Πρόεδρε από μια πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζει μια πολιτική της Ευρώπης φρούριο και από την άλλη πλευρά να πολλαπλασιάζονται οι επεμβάσεις και παρεμβάσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε μιλάμε για Αφγανιστάν, Πακιστάν, Αφρική, οποιασδήποτε χώρες. Λοιπόν, όσο υπάρχει αυτή η επεμβατική πολιτική θα οξύνεται το πρόβλημα της μετανάστευσης. Τρίτο ζήτημα. Μιλάω για την Ελλάδα. Απαράδεκτο το καθεστώς Απαράδεκτο από κάθε άποψη. Μιλάτε κύριε εισηγητά για το ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κατασταλτικές ε, πολιτικές. Συμφωνούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν φράχτες ενάντια στους μετανάστες όπως ξέρετε. Υπάρχει Frontex που ε, κυνηγάει τους μετανάστες. Δεν έχουν δικαιώματα οι μετανάστες. Καθόλου. Και είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά άλλα τέτοια ζητήματα. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτή την έκθεση. Θα κάνουμε τροπολογίες βεβαίως, αλλά η τελική μας τοποθέτηση θα εξαρτηθεί από το συνολικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Well, Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Θεοχάρους έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση του κυρίου Προβέρα είναι πολύπλευρη και ιδιαίτερα σημαντική και δεν πρέπει να ειδωθεί ότι από μόνη της θα πρέπει να δώσει λύσεις και απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι πάρα πολλά παράπλευρα θέματα τα οποία αναπτύχθησαν από τους συναδέλφους έχουν φυγεί και άλλος πως μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σωστά επισημαίνεται ότι η αστάθεια είναι ο κύριος λόγος ο οποίος οθεί τους πληθυσμούς να μετακινούνται προς τις πιο πλούσιες ας πούμε περιοχές αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την αστάθεια που προκαλείται στις χώρες υποδοχής γι' αυτό νομίζω ότι εμείς τουλάχιστον του μεσογειακού νότου που δεχόμαστε τους κραδασμούς αυτής της αστάθειας πρέπει να σας μεταφέρουμε και την κοινωνική εξέγερση που παρατηρείται αυτή τη στιγμή χωρίς αυτό να σημαίνει οτιδήποτε το ρατσιστικό. Ε, άρα το ζητούμενο είναι να ελέγξουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα κρατώντας τους ανθρώπους στις χώρες τους και εκείνοι που πραγματικά έχουν ανάγκη δεν νοιάζονται αν είναι ανθρωπιστική βοήθεια ή αναπτυξιακή βοήθεια. Σημασία έχει όμως εμείς να στοχεύσουμε την ε, βοήθεια ούτως ώστε να μπορούμε να τους κρατήσουμε ε, με τη θέλησή τους στη χώρα τους και να μπορούν να προκόψουν. Αυτό θα δώσει και στους ευρωπαϊκούς λαούς την αίσθηση ότι πραγματικά προλαμβάνοντας την αστάθεια μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρουν σωστά δαπανώντας κάποια, βοήθεια προς τους, αυτούς που την χρειάζονται. Επιπλέον πρέπει να επισημάνουμε και την ανάγκη για την ισομερή κάλυψη όλων των αναγκών που προκύπτουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μη ελεγχόμενη μετανάστευση. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Άννα. Για ένα λεπτό, Άννα, όχι δύο, ένα. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Προβέρα, τον ε, εισηγητή, που προσπάθησε να κάνει κάτι πολύ δύσκολο, δηλαδή να καταθέσει ε, σειρά στοιχείων. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα με τα οποία συμφωνώ, αντίστοιχα όμως και πράγματα με τα οποία δεν είναι ότι δεν, συμφωνώ, αλλά η πρακτική μας έχει αποδείξει το αντίθετο και νομίζω ότι για τη Μεσόγειο, για τη Βόρεια Αφρική ε, έχουμε τσεκάρει επανειλημμένα τις ε, δυνατότητές μας. Έχουμε δει ότι οποτεδήποτε έχουμε κάνει λάθος, οποτεδήποτε έχουμε πάρει μια λάθος απόφαση, στην ουσία ε, αυτό έχει γίνει μπούμεραγκ, έχει γυρίσει πάνω μας. Ε, ας πούμε η αιρεσιμότητα στη Συμφωνία Κοτονού ξέρουμε πάρα πολύ καλά που οδήγησε θα τελειώσω λέγοντας ότι ε, για το Μνημόνιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Λιβύης. Ε, στην ουσία το πρόβλημα εκεί είναι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και στη Λιβύη ακόμα και νομίζω ότι είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε τον ρόλο των ε, γυναικών ε, καθώς επίσης ε, και τις καταχρήσεις των οποίων, τις οποίες υφίστανται κυρίως οι γυναίκες και τα παιδιά αλλά γενικότερα οι μετανάστες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκουγιαβέρ για δύο λεπτά εσείς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Δύο σημεία τα οποία νομίζω ότι μπορούμε να αναφέρουμε. Σημείο 9 σχετικά με την ε, κυβερνητική διάσκεψη του UFM. Ε, η ύπατη εκπρόσωπος ασχολείται με το θέμα αυτό όσον αφορά δηλαδή, τις διαπραγματεύσεις, την επιχειρηματολογία ε, που σχετίζεται με την ε, μετανάστευση αλλά και με τα μέτρα πρόληψης και φυσικά με μέτρα καταπολέμησης του τράφικινγκ ας πούμε, συγκεκριμένων δηλαδή δράσεων. Επίσης, αναθεώρηση EMP θα εγκριθεί από την ε, Κομισιόν την 20η Φεβρουαρίου και εκεί θα λάβουμε υπόψη όλα αυτά που λέτε εσείς εδώ. Τελευταίο σημείο, η εντολή της ε, ε, Αντιπρόεδρου της Επιτροπής ΥΠΑ του εκπροσώπου σχετικά με όλα τα στοιχεία της πολιτικής ε, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα οποία θα πρέπει να είναι συνεκτικά και λέω θα πρέπει να περιλαμβάνουν και θέματα ανθρωπιστικά και θέματα οικονομικά και θέματα ε, πολιτικά ή αναπτυξιακά. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μαζί και με τα νέα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Προβέρα, έχετε το λόγο. Μου ζήτησε ο πρόεδρο ε, να σχολιάσω λακωνικά. Ευχαριστώ πολύ όλους τους παρεμβαίνοντε. Ε, συνάδελφε Γκόμες. Εγώ δεν προτείνω πολιτική, εγώ ζητώ ε, να σκεφτούμε, να αναρωτηθούμε όλοι μαζί, όλες οι πολιτικές ομάδες για την πολιτική μετανάστευση, αλλά στα πλαίσια μιας ευρύτερης πολιτικής ανάπτυξης. η αναπτυξιακή πολιτική, η πολιτική συνεργασία, η οικονομική βοήθεια δεν μπορούν από μόνα τους να κάνουν τίποτα. Ξέρουμε, έχουμε δει και στο παρελθόν περιπτώσεις όπου ε, μπορούσαμε να βοηθήσουμε, ξεκινήσαμε με προγράμματα και μετά η πολιτική αστάθεια, πόλεμοι κτλ. εξουδετερώσαν οποιαδήποτε προσπάθεια. Συνάδελφε Σάκε, ε, ναι βεβαίως αγαπητοί συνάδελφοι έχετε δίκιο. Ε, εγώ συμμερίζομαι την άποψή σας για το brain drain Βεβαίω, Βεβαίως εμείς μπορεί να θέλουμε νέους ε, έξοχους ε, ε, ερευνητές ή εξαιρετικούς επιστήμονες αλλά στην ουσία εμείς παίρνουμε κάθε δυνατότητα ανάπτυξης από χώρες του τρίτου κόσμου. Μοντάλτο, πολιτική εξωτερική δράση. Ναι, βεβαίω, οπωσδήποτε, οποιαδήποτε απόφαση για την γενική μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να συμβαδίζει με την εξωτερική πολιτική, έτσι ώστε οι λύσει που προτείνονται να είναι αποτελεσματικέ. Ένα είναι βέβαιο, ότι στο παρελθόν είχαμε σημαντικότατε αποτυχίε, παταγώδει αποτυχίε, από τι οποίε πρέπει να μάθουμε ε, τι δεν πήγε καλά, έτσι ώστε να τι αποφύγουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Να σα υπενθυμίσω ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι η 8η Φεβρουαρίου 2011 στι 12 το μεσημέρι και θα ξανασυζητήσουμε το ζήτημα αυτό ξανά στις 16 Μαρτίου. Πολύ γρήγορα προχωράμε στο επόμενο θέμα που είναι πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου. Να ζητήσω από τον κύριο Τάνοκ, ο οποίος είναι εισηγητής, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερα στη γραμματεία ε, της Επιτροπής μας που με βοήθησε πολύ για τη σύνταξη της έκθεσης αλλά και όλους τους κοιόδης εισηγητές με τους οποίους συναντήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα. Χάρη σε αυτούς ε, είναι αρκετά ομαλή θα έλεγα, ίσως από τις πιο εύκολες εκθέσεις που είχα να διαχειριστώ ε, τα χρόνια τα οποία είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρά τη σχετική αυτή ευκολία, ωστόσο, έλαβα 76 τροπολογίε, οι οποίε καλύπτουν του περισσότερου τομεί. Προσπάθησα σε συνεννόηση και με τους και όσοι όλους τους συνάντησα από τις βασικές πολιτικές ομάδες να καταλήξω σε κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις. Είναι 8 τον αριθμό, φαντάζομαι τις έχετε και έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, 2-3 βελτίωση δικαιωμάτων μειονοτήτων, 4-5 ε, ε, την οικιακή βία, τη βία κατά των γυναικών, ε, LTGP κοινότητες, εσωτερικώς εκτοπισθέντες, Ρωμά ε, και κάποιοι Αιγύπτιοι οι οποίοι έρχονται κυρίως στο Κωσυφοπαίδιο και κάποια άλλα θέματα, παραδείγματο χάρη ότι χρειάζονται εν γέννη περισσότεροι πόροι για το δικαστικό σύστημα, την ανεξαρτησία των δικαστικών, την εποπτεία, τον έλεγχο ε, του Κοινοβουλίου. Θα συναντηθώ με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς ε, για την ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών. Θα πρέπει επίσης και το Σύνταγμα του Μαυροβουνίου σε σχέση με τις εκλογές, στη Συμβαστική 1 βλέπουμε τις σχετικές προτάσεις και έχουμε και τη Συμβαστική 2 για κάποιους αξιωματούχους. Εγώ πρέπει να σας πω ότι σε μια πολύ μικρή χώρα 600 περίπου χιλιάδες κάτοικοι, ε, είναι πρόκληση ε, να μην υπάρξει κάποιο είδου σύγκρουση συμφερόντων, γιατί οι θύνοντες, ε, η άρχουσα τάξη δεν είναι και τόσο πολύ άριθμοι και επικαλύπτονται στις διάφορες αρμοδιότητες και θέσεις που έχουν. Επίσης, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, 7η προστασία δημοσιογράφων και 8η συμβαστική, παράγραφο 21. Την έχω τροποποιήσει για να έχουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες στον τομέα του περιβάλλοντος, φράγματα υδροελεκτρικά, κάτι που θα βοηθήσει να υπάρχει διαφοροποίηση της οικονομίας του Μαυροβουνίου, που είναι αρκετά μικρή κλίμακα και εξαρτάται υπερβολικά από τον τουρισμό. Νομίζω ότι είπα πολλά, είπα αρκετά και θα ήθελα να ακούσω και τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι. Θα ψηφίσουμε όμω στις 10 Φεβρουαρίου. Well, thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάνοκ. 1,5 λεπτό έχετε, κύριε Βουλευτά. Ίσως να μην τα χρειαστώ. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί ήταν πολύ καλή δουλειά του. Η έκθεση, για την πρόοδο, η έκθεση πρόοδο μάλλον για το Μαυροβούνιο δείχνει μια θετική γενικά στάση του Κοινοβουλίου προς τη χώρα αυτή. Η πρόοδος του Μαυροβουνίου ως προς ε, την προσχώρηση μέχρι στιγμής υπήρξε, θα έλεγα, λίγο πολύ ομαλή. Και αυτό υπογραμμίζεται και σε ολόκληρη την έκθεση. Τώρα, πού είναι οι βασικές ανησυχίες κατά την προσωπική μου άποψη. Διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα. Παραμένουν σημαντικά προβλήματα στο Μαυροβούνιο και η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει πολλές, πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες. Επίσης, η εκλογική νομοθεσία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κανόνες, αλλά και με το Σύνταγμα του Μαυροβουνίου. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει έναν πιο ισχυρό εποπτικό ρόλο ε, έναντι της κυβέρνησης. Επίσης, ευρύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στι διαδικασίε νομοθετικέ αλλά και τι συμβουλευτικέ, ιδίω ό,τι αφορά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το Μαυροβούνιο έχει να ε, εκπληρώσει και τα άλλα ορόσημα, τους άλλους σταθμούς που προβλέπονται από την Κομισιόν για να πληρωθούν ενταξιακές διαπραγματεύσεις, κάτι που ελπίζω να γίνει σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Μπρισάτζιτς. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους. Θεωρώ ότι ήταν καλή και ισορροπημένη η έκθεση την οποία κατήρθησε ο εισηγητής. Υποστηρίζω όμως και την κριτική που άσκησε ο κ. Κούκαν. Νομίζω ότι οι συμβιβασμοί του οποίου πετύχαμε ενισχύουν το κείμενο και θα ήθελα να πω ότι το ΕΛΚ υποστηρίζει όλες τις, ε, όλες τις συμβαστικές προτάσεις. Ακόμα και των σοσιαλιστών τις ε, τροπολογίες υποστηρίζω. Σχεδόν όλες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνο για την καλή δουλειά που έκανε και το γεγονός, για το γεγονός ότι αποδέχτηκε τροπολογίες από διάφορες ομάδες, όχι μόνο από τη δική μου ομάδα, για θέματα που ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για μας. Νομίζω ότι το κείμενο περιλαμβάνει πλέον όλα τα σημαντικά στοιχεία ως προς την πρόοδο του Μαυροβουνίου με καλή διατύπωση που διασαφηνίζει ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι θα πρέπει να κάνει στο μέλλον το Μαυροβούνιο. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και αυτά που είπε ο κ. Στάνοκ σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη διαφθορά στο θέμα των μειονοτήτων, των μέσων. Όλα αυτά είναι θέματα δημόσια διοίκηση, θέματα που περιλαμβάνονται στο κείμενο και τα εκτιμώ. Και εκτιμώ και το πνεύμα συνεργασία που έδειξε ο κύριος Τάνοκ. Θα ήθελα να σχολιάσω τρεις ε, τροπολογίε. Η πρώτη είναι και την, αναφερθε... την αναφέρετε και εσείς ε, κύριε Τάνοκ, είναι 38 για τις μειονότητες, για τους Ρωμά και το καθεξής. Τους Ασκαλούς και τους Αιγυπτίους ζητάτε την ενίσχυση της εφαρμογής των νόμων που υπάρχουν. Ελπίζω να αλλάξετε την ε, γνώμη σας, γιατί όπως ξέρετε είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή. Μπορεί να υπάρχουν οι νόμοι, αλλά να μην εφαρμόζονται. Άρα θα θέλαμε να αλλάξετε την γνώμη σας και ίσως να υπερψηφίσουν και οι συνάδελφοι την τροπολογία μας και άλλη μία τροπολογία. Η 73 για τη συμφωνία, για τη δημιουργία ε, μεταξύ ε, Ιταλίας και Μαυροβουνίου για δίωδο ενέργειας, για αγωγό ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξέτασε την έκθεση, δήλωσε ότι της αρέσει ο τρόπος που διατυπώνεται η τροπολογία αυτή. Ελπίζω να την υπερψηφίσουν οι συνάδελφοι. Τελευταίο στοιχείο. Ναι, τελευταίο, τελευταίο, τελευταίο στοιχείο. Για την κατάσταση την υδροηλεκτρική. Συμφωνώ με όσα είπε ο κύριος Τάνοκ για την ανάγκη να υπάρξει ποικιλία γνωρίζοντας ότι το Μαυροβούνιο έχει και την μεγαλύτερη πηγή μάλλον ενέργεια στο Μαυροβούνιο είναι η υδροελεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, υπάρχει το θέμα το κατά πόσο θα ακολουθήσουμε το συμβιβασμό ή θα υποβάλουμε προφορική τροπολογία λίγο πιο ε, έντονη ως προς τη διατύπωση για να ζητήσουμε θα ζητήσουμε μια καλή οικολογική εκτίμηση. Ελπίζω να υπάρχει όμως και άλλο περιθώριο πραγμάτευσης μέχρι την... Ε, ε, κύριε Σκουντής, ένα λεπτό. Ενάμιση λεπτό, κύριε Σκουντής. Πρόεδρε, η έκθεση του συναδέλφου πράγματι είναι ισορροπημένη. Έχει κάνει σοβαρή δουλειά. Άλλωστε δεν είχε και μεγάλες δυσκολίες όπως και ο ίδιος ομολόγησε. Αυτό σημαίνει ότι στο στάδιο και στο κομμάτι που καταγράφει τα προβλήματα και τις πρόοδους που έχει γίνει δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Επίσης ε, είμαστε γενικά σύμφωνοι με τις ε, συνενετικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, θα πω που διαφωνούμε και βεβαίως με την προφορική τροπολογία που κατέθεσαν οι πράσινοι. Δεν συμφωνούμε κύριε Πρόεδρε και κύριε Σιγητά με τη συνενετική τροπολογία όπου εμφανίζεται για άλλη μια φορά το γνωστό πρόβλημα. Για να ενταχθεί μια χώρα, μια χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, επί της αρχής η ομάδα μας γενικά λέει ναι μπορεί να ενταχθεί εφόσον ο λαός το επιθυμεί τίθενται μια σειρά δεσμεύσεις που έχουν να κάνουν με την επιβολή νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Μιλάμε για ιδιωτικοποίησεις, μιλάμε ουσιαστικά για διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών, μιλάμε για εφαρμογή της πολιτικής της Μπολόνια. Αυτά δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Και δεν μας βρίσκουν σύμφωνος όχι μόνο επί της αρχής δεύτερο διότι περιορίζουν τη δυνατότητα επιλογής πολιτικής και οικονομικής πολιτικής μιας χώρας και τρίτο κινούνται στο πολύ λαθεμένο σχήμα ότι οι η ελευθερία των αγορών φέρνει και δημοκρατία, φέρνει και πρόοδο στο επίπεδο των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Αυτό το σχήμα έχει αποτύχει. Επομένως είναι ατυχές, αν δεν είναι λαθεμένο, να επιμένουμε προκειμένου να ενταχθεί μια χώρα να της υπαγορεύσουμε όλες αυτές τις πλευρές της πολιτικής την τελική μας στάση θα την καθορίσουμε από το πώς θα εξελιχθεί το τελικό κείμενο. Ευχαριστώ. Thank you very much. For one minute, Mr. please. Κατσίν, για ένα λεπτό. Α, όχι, ήταν ναι, ναι, Βάγγελ, Βάγγελ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξακολουθούμε να είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα στο Κοινοβούλιο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να συνταχθώ με τους συναδέλφους που εξεθίασαν την εργασία του εισηγητού Τάνοκ. Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί του και εμείς ετοιμάσαμε και έξι τροπολογίες, οχτώ τροπολογίες ε, με τις οποίες συμφωνήσαμε όλοι και δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να προσθέσω. Θα ήθελα απλώς να υπογραμμίσω ότι ακόμα περιμένουμε. τα αποτελέσματα της Επιτροπής που ξεκίνησε την εργασία της πριν από μερικά χρόνια σχετικά με τα αντικρουόμενα συμφέροντα ε, και νομίζω ότι θα πρέπει ε, όντως να ενταθεί η προσπάθεια καταπολέμησης διαφθοράς, μια και η διαφθορά ακόμα καλά κρατεί στη χώρα αυτή. Κάτι άλλο που ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι θα πρέπει να ε, υπάρξει περαιτέρω προσπάθεια ε, έτσι ώστε να είναι καλύτερη η ελευθεροτυπία, η ελευθερία των μέσων ε, ενημέρωσης γιατί είναι κρίμα, είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα, μια μικρή όμορφη χώρα ε, η οποία καλό θα ήταν να, γίνει πλήρες μέλος. Τώρα ένα λεπτό κύριος Κατσίνου. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. είναι πολύ θετικό απέναντι σε αυτή τη μικρή χώρα που έρχεται όλο και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι καλό θα ήταν σε μια προφορική τροπολογία να ενθαρρύνουμε και τον ε, νέο Πρωθυπουργό που ανέλαβε καθήκοντα και συναντήθηκε και με τον ε, Σότι Μέρα ανάληψη των καθηκόντων του. Αν ε, φέρατε κύριε Τάνοκ ότι θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα κάπω ασυνήθιστο ε, πρόβλημα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας ε, έχει χτίσει μια εκκλησία. Χρησιμοποίησε όμως ελικόπτερα του πρώην Κοσλαβικού στρατού και τώρα ζητείται η κατεδάφιση, η απομάκρυνση αυτού του ναού. και μάλιστα έχει αφοριστεί, έχει καταραστεί τον ε, πρόεδρο εκεί. Δεν είναι αυτός ε, ο τρόπος με τον οποίο κανονικά έπρεπε να επιλύονται ζητήματα τον 21ο αιώνα. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει κάπως να πέσουν οι τόνοι Έχουμε και κάποιες ε, ποινικέ διαδικασίες ε, που θα ε, επισύρουν έτσι και με κάποια αρνητική προσοχή. Θα ήθελα κύριε Τάνοκ να κάνετε ό,τι μπορείτε. ώστε το παρελθόν να μην υποσκάπτει το παρόν και το μέλλον. Καλώς ήρθατε στα Βαλκάνια, λέει ο Πρόεδρος. Ε, κύριε Τάνοκ, έχετε πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι παρά το προειδοποιητικό ε, σήμα να προσέξω γιατί θα αναλάμβω μια έκθεση για τα Δυτικά Βαλκάνια τελικά βλέπω ότι υπάρχει σχετική συνένεση νομίζω ότι η Γκουε παραπονέθηκε μόνο για τη λέξη ιδιωτικοποίηση αυτό είναι αρκετά αξιοσημείωτο Λοιπόν, α αναφέρω σύντομα, σύντομα κάποια πράγματα. Κύρια Τσέκα για την παράγραφο 38. Κοιτάξτε, θα εξετάσω και πάλι τη διατύπωση. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο προσβλητική. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς ε, ποια ήταν η λογική που με έκανε να εκφραστώ έτσι, αλλά θα έρθω σε επαφή με τους συναδέλφου και θα επανέλθω. Νομίζω όμως ότι μάλλον μπορούμε να υποχωρήσουμε και να δεχθούμε το έτοιμά σας. Σε ό,τι αφορά το 73, ενημερώθηκα ότι είναι παροχημένη αυτή η τροπολογία υπήρξε δημοσίευση από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου, θα το ελέγξω όμως και θα στείλω email σε περίπτωση που είναι πλέον περιττή αυτή η τροπολογία γιατί δεν συμβαδίζει, δεν είναι επικαιροποιημένη αν θέλετε, αλλά θέλω κάποιες διευκρινήσεις. Θα υποστηρίξω την ε, προφορική τροπολογία ε, για την συμβιβαστική τροπολογία της παραγράφου 21. Για τον κύριο Κατσίν τώρα. Θα είμαι υπέρ κάθε προφορικής τροπολογίας για το ρόλο του νέου Πρωθυπουργού από ό,τι καταλαβαίνω, ένα ιδιαίτερα ταλαντούχο νέο. Υπήρξε υπουργό οικονομικών στην Ποντγκόριτσα, τον είχα συναντήσει για λίγο. Και νομίζω ότι δεν κάνω λάθο αν πω ότι αναφέρουμε το ότι το Μαυροβούνιο πλέον έχει το καθεστώς επίσημη υποψήφια χώρας, στι αιτιολογικές σκέψει δεν αναφέρεται και πρέπει κάπου να το προσθέσουμε. Είναι μια τεχνικής ε, φύσεως τροπολογία αυτή. Τώρα σε ό,τι αφορά το ρόλο του νέου Πρωθυπουργού και για τα, αυτά τα κλησιαστικά ζητήματα, δυστυχώς δεν το γνωρίζω αυτό που είπατε, πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο αν και διαβάζω ε, τι γίνεται εκεί, αλλά δεν γνωρίζω και τη γλώσσα για να ε, έχω όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Αν έχετε την καλοσύνη να με ενημερώσετε, θα το εκτιμήσω όλος ιδιαίτερος. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ε, τελειώσουμε, κλείσουμε τη συζήτηση, να σας πω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την 10η Φεβρουαρίου αποφασίσαμε ότι η συνέχιση της συνεδρίασης θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω όσους δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην αίθουσα να εγκαταλείψουν την αίθουσα αυτή. The meeting is